Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την συνεδρίαση σήμερα. Δεν θέλω να προχωρήσω με τις ανακοινώσεις του Προέδρου, αλλά θέλω να πω ότι όλοι χαιρόμαστε για τη συμφωνία της Πριστίνας και πιστεύουμε η συμφωνία της Πριστίνας με το Βελιγράδι συνήφθη και θα συζητήσουμε αύριο τη συμφωνία αυτή διότι είναι ένα σημαντικό γεγονός για την περαιτέρω διαδικασία της ανάπτυξης των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Και έτσι προχωρούμε κατευθείαν στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Υπάρχει καμία αντίρρηση, παρατήρηση στα πρακτικά, αν, αν κάποιος τα διάβασε δηλαδή. Ωραία, δεν υπάρχει τίποτα. Στο 3 προχωρούμε λοιπόν στο 4 με ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τον εξοχότατο Μοχάμετ Αλ Ίζα, και θα συζητήσουμε τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος της Σαουδικής Αραβίας. Ένα, είχαμε ήδη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιστεύω ότι το θέμα αυτό έχει εξέχουσα σημασία και λόγω της ουσίας και λόγω της σημασίας της Σαουδικής Αραβίας. Ξέρουμε ότι η Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα, τα κράτη του Αραβικού κόλπου, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή αυτή του κόσμου. Συνδέονται τα θέματα αυτά και με τη Συρία και με την Αίγυπτο και ε, επίσης γίνονται προσπάθειες κωδικοποίησης ε, του Ισλαμικού νόμου, τη Σαρία και θέλουμε να συνδέσουμε με όλα τα θέματα αυτά και τις, ε, τους στόχους μας για το κράτος δικαίου, τις φιλελεύθερες πτυχές, ερμηνείες κλπ. Και γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω τη συζήτηση. Έχουμε βεβαίως και ερωτήσεις που αφορούν τη θανατική ποινή και άλλα συναφή θέματα. Αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με το Ισλαμικό δίκαιο, αλλά έχουν επιπτώσεις στο όλο πλαίσιο του δικαίου και εάν το δίκαιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, διαφέρει ή συνάδει με, το διεθνές δίκαιο. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα λοιπόν προς συζήτηση και θα ήθελα να δώσω θα δώσω το λόγο στον εξοχότατο Υπουργό. Στο όνομα του πολύ, ε, πολύ ε, ελεήμονος και πολύ εύστοχου Θεού, χαίρομαι που είμαι μαζί σας σήμερα. Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή, στην οποία μετέχουν σήμερα εκπρόσωποι ε, στην οποία μετέχουμε σήμερα αντιπροσωπεύει την ενίσχυση της συνεργασίας μας μεταξύ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στην Σαουδική Αραβία δηλαδή είναι ένα θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι το δικαστικό σύστημα στην Σαουδική Αραβία ε, δείχνει ότι χρειάζεται μια νέα νομοθεσία που ρυθμίζει την ε, δικαστική εξουσία και αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. δίνοντας την δικαιοσύνη στη χώρα μου όλα τα μέσα που θα της επιτρέψουν να έχει μια μεγαλύτερη αμεροληψία και ανεξαρτησία. Η νομοθεσία για τις ε, δικαστικές αρχές που είναι πολύ καινούργια νομοθεσία μεταρρύθμισε βαθιά πολλές διατάξεις ε, της υφιστάμενης νομοθεσίας. Βασίζεται δε στις πιο σύγχρονες αρχές της δικαιοσύνης που παρέχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία, και ουδετερότητα στη δικαιοσύνη, ενώ προβλέπει διατάξεις που επιβεβαιώνουν την αρχή της δημόσιας, της δημοσιότητας της δίκης, κάτι που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, η ΜΕΔΑΠΑ και αλλοδαπά να γνωρίζουν την ε, επακροατήριο διαδικασία μιας δίκης, να παρακολουθούν τη διαδικασία αυτή και τούτο χωρίς επιφύλαξη και χωρίς εξαίρεση. Για μας η δικαιοσύνη είναι τελείως ανοιχτή, διάφανη. Τα μέσα ενημέρωσης στην ε, Σαουδική Αραβία ιδίως ε, μεταδίδουν ακροαματικές διαδικασίες με αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Μεταξύ των εγγύσεων που προσφέρει η δικαιοσύνη της χώρας μου υπάρχει και ο νόμος που αφορά στην αστική δικονομία και ένας άλλος νόμος που αφορά στην ποινική δικονομία. Η νομοθεσία αυτή βασίζεται στις πιο σύγχρονες αρχές και δράσεις των ε, διαφόρων χωρών του κόσμου. Η βάση της δικαιοσύνη και του δικαστικού συστήματος στη Σαουδική Αραβία ε, στηρίζεται και συμμορφώνεται με αυτό που γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όσο αφορά τις γενικές αρχές, η φιλοσοφία η δικαστική φιλοσοφία μας δεν αντιβαίνει ουδόλως στην δικαστική φιλοσοφία που υπάρχει ε, σε άλλες χώρες του κόσμου είτε μιλάμε για την αστική δικαιοσύνη, είτε για την ποινική, είτε για το εμπορικό δίκαιο. Στη Σαουδική Αραβία αυτό που θεωρούμε σημαντικότερο είναι να μην υπάρξει αντίφαση με τα συνταγματικά κείμενα που εμπνέονται από το κανονικό μουσουλμανικό δίκαιο, την Σαρία. Η Σαρία διέπει όλες τις δικαστικές διατάξεις στην χώρα μου, αλλά με εξαιρετικά λιτό τρόπο. Υπάρχει μια διακριτική, πολύ σημαντική διακριτική εξουσία που έχει ο δικαστής, η δικαιοσύνη. Ο δικαστής λοιπόν έχει κάθε περιθώριο ερμηνείας της Σαρία και να αντλήσει την απόφαση, να στηρίξει την απόφασή του είτε σε προγειονέστερη νομολογία είτε σε δική του ερμηνεία του νόμου. Είναι λοιπόν το σύστημά μας ένα νομολογιακό κατά βάση σύστημα. Επίσης έχουμε νόμους που εκδίδει ο νομοθέτης και που αφορούν την στενή ενία απονομή της δικαιοσύνης. Στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχουν ε, δικαστήρια που είτε δικαστήρια ασφαλείας του κράτους είτε ε, δικαστήρια που αντιμετωπίζουν με έκτακτο τρόπο τα, ε, τα γεγονότα. Όποιος ε, θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη μπορεί να προσφύγει με απόλυτη ελευθερία μέσω των τακτικών δικαστηρίων. Αυτό ακριβώς ε, είναι, αυτό ακριβώς στηρίζεται στη βούλησή μας να απονείμεται δικαιοσύνη σε όλους δικαιοσύνη καλύπτεται απόλυτα από το κράτος με την εξαίρεση των αμοιβών των ε, δικηγόρων. Για μας η δικαιοσύνη δεν έχει τίμημα, αποτελεί ευθύνη του κράτους έναντι όλων. Το κράτος λοιπόν καλύπτει όλες τις δαπάνες δικαιοσύνης, όλες τις δικαστικές δαπάνες για όλους. Ομοίως, διευρύναμε την αρχή της ε, δικαστικής ειδικότητα. Υπάρχουν δικαστήρια κοινού δικαίου, δικαστήρια εμπορικά, υπάρχουν ποινικά δικαστήρια, δικαστήρια οικογενειακής προσωπικής κατάστασης, εργατικά δικαστήρια Και μπορούμε επίσης εκ του νόμου να δημιουργήσουμε και άλλα δικαστήρια ανάλογα με την ανάγκη. Βεβαίως ε, υπάρχει πάντα το επίπεδο της έφεσης και εκεί υπάρχει εξειδίκευση κατηγορία και υπάρχει και ένα ανώτατο δικαστήριο καθώς και ένα ανώτατο διοικητικό δικαστήριο για την διοικητική δικαιοσύνη. αυτό που στη χώρα μας αποκαλούσαμε Συμβούλιο Επικρατείας στην Ευρώπη. Οι αρχές τώρα που βλέπουν την, τη δικαιοσύνη στην Σαουδική Αραβία, οι αρχές αυτές είναι αυτονόητο, σέβονται όλες τις ε, διεθνείς ε, συμβάσεις, συνθήκες, συμφωνίες και νομικά κείμενα στα οποία, των οποίων είναι συμβαλόμενο μέρος η Σαουδική Αραβία. Το δικαστικό μας σύστημα σέβεται επίσης ε, την αλλοδαπή νομολογία και τα διαιτητικά, τις διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν στο βασίλειο. Και τούτο βάσει διμερών, πολυτερών ή πολυ, πολυμερών συγγνώμη, ή αμοιβαίων συμβάσεων που ισχύουν. Τα δικαστήρια του Βασιλείου της Αδικής Αραβίας έχουν ήδη γνωμοδοτήσει ζητώντας για την υλοποίηση μιας σειράς ε, αλλοδαπών αποφάσεων, αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων. Μεταξύ των άλλων αρχών στις οποίες ε, βασίζεται η δικαιοσύνη μας είναι ο σεβασμός ε, της ε, ελευθερίας της γνώμης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Την η ελευθερία έκφρασης γνώμης κατά την άποψή μας διακρίνει μεταξύ της έννοιας της ελευθερίας και της αταξίας ή του χάους. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ελευθερία και το χάος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η ελευθερία της γνώμης ε, επιτρέπει να ε, δεχτούμε δημιουργία αναταραχής ή την διάδοση δηλητηριωδών ιδεών. Επιτρέπουμε σε όλους να εκφράζονται εφόσον δεν επηρεάζεται η ελευθερία του άλλου και δεν θίγει τη δημόσια τάξη. Τα δικαστήρια μας έχουν εκδώσει πάρα πολλές αποφάσεις και γνωμοτήσεις που συνάδουν με την αρχή αυτή. Όπως σας είπα, συνολικά σεβόμαστε τις αποφάσεις των αλλοδαπών διαιτητικών ε, δικαστηρίων και τα δικαστήρια μας δεν μπαίνουν στην ουσία των σχετικών υποθέσεων εφόσον δεν αντιβαίνουν οι αποφάσεις στις αρχές του κράτους. Οι μόνες παρεμβάσεις των δικαστηρίων μπορούν να αφορούν μόνο δικονομικά ζητήματα. Η δικαιοσύνη της Σαουδικής Αραβίας σέβεται επίσης τις οργανώσεις δικαιωμάτων την επιτρέπει μάλλον στις οργανώσεις δικαιωμάτων ανθρώπου να ασκούν τη δράση και υιοθετήσαμε μια σειρά εκθέσεων μη κυβερνητικών οργανισμών τόσο εθνικών όσο και διεθνών Και για να ε, ενεργοποιηθεί αυτή η αρχή της διαφάνειας που σας ε, ανέφερα προηγουμένως, προβλέψαμε ένα σύστημα υποστήριξης των ΜΚΟ που ε, ρυθμίζεται από μια εθνική δομή διαφάνειας και ακαιρεότητας. Η δομή αυτή αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό όλων των τοπικών και διεθνών ενώσεων και μη κυβερνικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. αυτή η δομή ακαιρεότητας και διαφάνειας συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με εθνικές και διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Πιστεύω ωστόσο ότι με αυτά που σας είπα έχετε μια γενική εικόνα της κατάστασης στη Σαουδική Αραβία. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για, την εισήγησή σας. Καλώς ορίζω και τον κύριο Φλόρενς, τον συνάδελφό μα από... Ε, και την ομάδα επισκεπτών του και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοχ Μπίλερ, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στο Κοινοβούλιο να ε, μας μιλήσετε. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Αύριο λοιπόν. Οπότε περιορίζουμε σήμερα σε δύο θέματα. Καταρχάς θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να υποβάλει μια ανέκτηση τον Ιούλιο στο Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη μεγάλη Ισλαμική χώρα η οποία δεν έχει επικυρώσει τις δύο νομικά δεσμευτικές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, αστικά δικαιώματα, τις δύο αυτές συμβάσεις. Θα ήθελα να μας πείτε εάν γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις μέσα στην κυβέρνησή σας για να ε, αναπτυχθεί ένας οδικός χάρτης προς την επικύρωση των συμβάσεων αυτών. Έχετε ήδη επικυρώσει τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων, τη σύμβαση κατά της διάκρισης εναντίον των γυναικών, αλλά έχετε μεγάλες επιφυλάξεις ως προς αυτές τις δύο που εκκρεμούν. Επίσης, ερωτώ, ε, θα αναπτύξει, έχετε καθοδόν μια διαδικασία που θα δώσει δυνατότητα άρσης αυτών των επιφυλάξεων. Όπως ξέρετε, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη όσον αφορά την κατάρριξη της θανατικής ποινής. Και στη Σαουδική Αραβία πολλά εγκλήματα, πολλά ποινικά αδικήματα επιφέρουν τη θανατική ε, ε, ποινή, όπως παραδείγματο χάρη ναρκωτικά, ε, μαγεία και άλλα εγκλήματα. Υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσετε προς ένα μορατόριο που θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την κατάργηση θανατικής ποινή. Και δεύτερον, στην περιοδική αναθεώρηση του ΟΗΕ, η Σαουδική Αραβία έχει προτείνει τον περιορισμό της, του πεδίου ισχύου της θανατικής ποινή ως ε, τιμωρία για ποινικά δικήματα. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε, να μας ενημερώσετε, ε, κατά, αν έχετε προχωρήσει στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογή. Τη της θανατικής ποινής. Η κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε σε εμά. να συζητήσουμε τα θέματα μας. Θα ήθελα ίσως και εγώ να αφήσω τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αυριανή συζήτηση, ε, τα θέματα των αλευθεριών, την εξαρτησία του δικαστικού σώματος και πώς εφαρμόζεται στη χώρα σας. Παραδείγματο χάρη ε, δεκάδες γυναίκες και παιδιά διαμαρτυρήθηκαν διότι δεν έχουν πρόσβαση ε, στους άντρες τους, στους συζύγους, στους πατέρες τους οι οποίοι βρίσκονται ε, στη φυλακή, είναι έγκλειστοι ενδεχομένω για τρομοκρατικά δικήματα. Ήθελε λοιπόν να ρωτήσω, α, επειδή υπάρχει και περιορισμό στη χρήση του Twitter, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών σας, αλλά όλα αυτά θα τα αφήσω για αύριο. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, του, και της δικονομίας και την ε, δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε γυναίκες ε, δικηγόρους και ακριβώς επειδή η Σαουδική Αραβία παίζει ένα σημαντικό ρόλο, άλλοτε θετικό, άλλοτε αρνητικό. Εγώ γύρισα σήμερα από τη Λιβύη που... και ξέρω το ρόλο που παίζεται στις ε, χώρες της ε, Αραβικής Άνοιξης. Ε, βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες οι οποίες χρηματοδοτούνται από τη Σαουδική Αραβία καταπιέζουν ε, το γυναικείο πληθυσμό. Ε, οι οποίες γυναίκες έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την Αραβική Άνοιξη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε να με ενημερώσετε τι γίνεται με το γυναικείο κίνημα στη χώρα σας. Στη Συρία ε, πιστεύω ότι χωρίς να το θέλετε, δηλαδή όχι σκόπιμα, αλλά όπλα διοχετεύονται στη Συρία και χρησιμοποιούνται είτε από παδού τη αλ ε, κατά έναν τρόπο τον οποίο δεν επιδιώξατε εσείς. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε την κατάσταση στο Μπαχρέιν διότι 70% του πληθυσμού αισθάνονται αποξενωμένοι, απομονωμένοι, από τα, στερημένοι από τα πολιτικά τους δικαιώματα και έγιναν διαδηλώσεις, απελάστηκαν, απε, απελάστησαν ε, ξένοι ε, δημοσιογράφοι. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση στο Μπαχρέιν. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ο πρόεδρος, η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Με τη σειρά μου θα ήθελα να συνεχίσω τις ερωτήσεις που έχουν θέσει ήδη οι κυρίες Λοχμπίλερ και Γκόμες. Θεωρώ ότι επέδειξε θάρρος ο κύριος υπουργό που προσήλθε ενώπιον μας για να μας εξηγήσει την προσπάθεια εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης στη χώρα του, που νομίζω ωστόσο ότι ο εξυγχρονισμός αυτός πρέπει να ικανοποιεί μια προϋπόθεση. Το δικαιικό σας σύστημα βασίζεται στη Σαρία. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Σαρία δεν προβλέπει ίσα δικαιώματα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Η κυρία Λόχ Μπίλερ ήδη μίλησε για μια συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών που ακόμα δεν έχετε υπογράψει. Εξακολουθούν εξακολουθεί δε να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Και αυτό για μας είναι πρόβλημα. Ρωτώ, διαρωτώ με μάλλον, γιατί δεν προδιαγράφει η νομοθεσία το τι θα πράξει η ε, δικαιοσύνη. Διότι επιβάλλονται νόμοι της Σαρία και σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Και αν δεν χωριστεί ο ρόλος της θρησκείας από την κρατική λειτουργία, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Γιατί δεν διαλέγεται ένα άλλο σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει αντικειμενικότητα απέναντι σε κάθε άνθρωπο στη χώρα σας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που εμφανιστήκατε ενώπιόν μας και μας απευθύνατε τα λόγια αυτά για ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε ότι μας απασχολεί έντονα. Ήδη προλαλήσατε, αναφέρθηκαν σε ορισμένα από τα θέματα που ήθελα να συζητήσω και εγώ μαζί σας, λέει η κυρία Νέιτς. Θέλω να σας θέσω το θέμα της θέσης των γυναικών στη σαουδική κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζει το δικαιικό σας σύστημα ή μάλλον το δικαιοδοτικό σας σύστημα. Είδαμε κάποια σημάδια κάποια αργής πρόοδου, αλλά τέλος πάντων πρόοδος είναι. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το πώς βλέπετε τις μελλοντικές εξελίξεις και εάν μου επιτρέπετε θα ήθελα να αναφερθώ, να σας παραπέμψω μάλλον, σε μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη στα αραβικά έθνη, που η έκθεση αυτή συντάχθηκε αποκλειστικά από Άραβες διανομένους και opinion leaders και η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για αυτό που αυτοί θεωρούν αργή ανάπτυξη, αν θέλετε αργή εξέλιξη σε διάφορες αραβικές κοινωνίες και βεβαίως αυτά ήταν πριν από την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Λοιπόν, ένας από τους σημαντικούς λόγους είναι ότι οι γυναίκες, δηλαδή το μισό της ανθρωπότητας, αποκλείονται από την κοινή ζωή. Και ο Κλοντ Λεβιστρός, γνωστός κοινωνιολόγος, που έφτασε μάλιστα την αξιοσέβαστη ηλικία των 101 ετών, έγραψε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι το γεγονός ότι σε ένα αριθμό κοινωνιών οι γυναίκες αποκλείονται από την δημόσια ζωή είναι ένας από τους λόγους της αργή τους εξέλιξης, αργής εκλέξης των κοινωνιών αυτών. Αυτά τα έγραφε στους θλιμμένους τροπικούς μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας κυρίες και κύριοι και χαίρο ε, που για τις ερωτήσεις σας ελπίζω οι απαντήσεις μου να είναι ικανοποιητικές. Για τα δύο σύμφωνα που αναφέρθηκαν η Σαουδική Αραβία και από την εθνική νομοθεσία και από τις συμβάσεις τις οποίες είναι συμβαλόμενο μέρος μεριμνά ώστε να υλοποιήσει τις περισσότερες από τις διατάξεις των δύο αυτών συμφώνων. Όταν ε, ενημερώθηκα για τα σύμφωνα αυτά, διαπίστωσα ότι οι περισσότερες διατάξεις που περιλαμβάνουν τα σύμφωνα αυτά ε, γίνονται σεβαστές από το βασίλειό μας. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις, ορισμένες διατάξεις των συμφώνων, δικαίωμα κάθε κράτους άλλωστε είναι αυτό, είναι τμήμα του διεθνούς δικαίου. Οι επιφυλάξεις, επιτρέπεται να, υποβάλλονται επιφυλάξεις σε διατάξεις. Και άλλωστε υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες διατάξεις των συμφώνων αυτών. Και εμείς ε, στη Σαουδική Αραβία θέλουμε να ασκήσουμε το δικαίωμα υποβολής επιφυλάξεων. Να σας λέω ότι η πλειοψηφία, οι περισσότερες διατάξεις των συμφώνων αυτών εφαρμόζονται στο εσωτερικό του βασιλείου. αν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα επιφυλάξεων στα δύο αυτά σύμφωνα που φύγουν κάποιους βουλευτές εδώ, ενημερώστε με σας παρακαλώ για να μπορέσω να σας εξηγήσω σε ατομικό επίπεδο τους λόγους. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι όλες οι επιφυλάξεις στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Τώρα, για τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων, την ΚΑΤ. Όπως και για την σύμβαση απαγόρευση των διακρίσεων κατά των γυναικών, εμείς επικυρώσαμε τις δύο αυτές συμβάσεις με επιφυλάξεις για κάθε διάταξη που αντιβαίνει σε μια συνταγματική αρχή του Βασιλείου. Δικαίωμά μας είναι αυτό, όπως κάθε άλλου κράτους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ωστόσο ότι οι αρχές αυτές αποτελούν απόσπαστο τμήμα του συντάγματος του Βασιλείου και δεν ε, νομίζω ότι οι επιφυλάξεις αυτές ε, έχουν βλάψει τις γυναίκες ε, της Σαουδικής Αραβίας και θα σου εξηγήσω. Για τη θανατική ποινή τώρα. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Επιτροπής σωστά υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία δεν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Εκατό χώρες την εφαρμόζουν. Υπάρχουν θεωρίες, φιλοσοφίες ε, που παρουσιάζουν, έχουν, πάνω, παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις. Όταν τόσο μπαίνουμε ε, στα ζητήματα αυτά, πρέπει να εφαρμόζουμε ένα κριτήριο λόγου, λογικής και να μην θεωρούμε να μην δρούμε κατά του δράστη του εγκλήματος με μεγαλύτερη φιλευσταχνία από ό,τι κατά του θύματος. Σε εμά η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και πολύ σπάνια. Όταν οι περιστάσεις του εγκλήματος είναι τέτοια, τόσο σοβαρές όταν υπάρχει για παράδειγμα προμελέτη, ε, φόνος, τότε η δικαιοσύνη επιβάλλει την θανατική ποινή, αλλά πρόκειται για κάτι πολύ σπάνιο. Ξέρω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν θεωρητικοί που πίστευαν ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια ότι η θανατική ποινή ήταν κάτι χρήσιμο για την κοινωνία. Εγώ κρίνω ότι εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία σε διεθνές επίπεδο για το θέμα της θανατικής ποινή, το θέμα παραμένει καθόλου ανοιχτό και νόμιμο. Επιπλέον, οι καταδικασμένοι σε θάνατο στους περασμένους αιώνες στην Ευρώπη καταδικάστηκαν βάσει ποιας λογικής των θεωρητικών, των φιλοσόφων κατόπιν. Ο δολοφόνος σε εποχή ειρήνης. Όταν δεν φωνεύεται ο ίδιος, τι δικαιοσύνη έχουμε. Και βέβαια πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της δολοφονίας εν ψυχρό σε καιρό ειρήνης και ενός μιας θανάτου, ενός θανάτου σε περίοδο πολέμου. Κατόπιν, για το δεύτερο, για τη δεύτερη ερώτησή σας, μιλήσατε για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Και για διαδηλώσεις γυναικών και παιδιών. Εγώ στη δουλειά μου ως Υπουργός Δικαιοσύνης διαπιστώνω ότι περισσότεροι από αυτούς που μετέχουν στις διαδηλώσεις αυτές ήταν ε, γυναίκες οι σύζυγοι των οποίων κατηγορούνται για τρομοκρατία. Άτομα δηλαδή που έλαβαν μέρος σε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά σαουδαραβικών ή αλλοδαπών στόχων. καλό το συνέστημα, αλλά πρέπει να έχουμε και ευθύνη. Και η ευθύνη μου είναι να εξασφαλίσω την ε, ασφάλεια και ακαιρεότητα των κατοίκων της χώρας μου. Οι διαδηλωτές αυτές, οι διαδηλώτριες αυτές ήθελαν την απελευθέρωση ατόμων τρομοκρατών που είχαν δικαστεί, καταδικαστεί Δεν είναι δυνατόν αυτό, το καταλαβαίνετε. Σεβόμαστε την ελευθερία έκφρασης. Όλοι έχετε, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν την ε, ελευθερία έκφρασης. Δεν υπάρχει εξαίρεση σε αυτό. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην ε, σαουδαραβική δικαιοσύνη. Προφανώς η γυναίκα έχει ρόλο στην κοινωνία μου και στη δικαιοσύνη της χώρας μου και τον διαδραματίζει απόλυτα. Σας καλώ να δείτε τι γίνεται στην πραγματικότητα της σαουδαραβικής κατάστασης πριν ε, και να μην στηρίζετε μόνο στις προκαταλήψεις σας. Η γυναίκα στην Σαουδική Αραβία μπορεί να ε, είναι δικηγόρος εδώ και 40 χρόνια. Εγώ ή ο ίδιος έχω υπογράψει την άδεια ε, γυναικών δικηγόρων, διότι στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ακόμα ε, δικηγορικοί σύλλογοι που τώρα εκδίδουν τις άδειες. Η γυναίκα σήμερα είναι ένα απόσπαστο τμήμα του δικαστικού σώματος ε, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως είπατε, το σύστημα, ε, όπως σας είπα, το σύστημα της χώρας μου στηρίζεται στο μουσουλμανικό κανονικό δίκαιο, την Σαρία. Πιστεύετε από ό,τι κατάλαβα ότι η Σαρία δεν εγγυάται πλήρη ισότητα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και δογμάτων του πληθυσμού. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η βασική αρχή της Σαρία είναι η απαγόρευση κάθε διάκρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως της θρησκείας, του χρώματος ή της φυλής τους. Καμία απόφαση δικαστηρίου στην Σαουδική Αραβία δεν εκδόθηκε βάσει εθνοτικής φιλετικής φιλετικής ή θρησκευτική διάκρισης. Αυτό απαγορεύεται. Η βασική αρχή της δικαιοσύνης μας είναι η αυστηρή ισότητα μεταξύ ε, πολιτών και κατοίκων της δικαιοσυνης μας ειναι η αυστηρη ισοτητα μεταξυ πολιτων και κατοικων της χωρας Και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να υπογραμμίσω ότι οι διατάξεις του κανονικού δικαίου του Ισλάμ που περιλαμβάνουν διαφορετικές ρυθμίσεις είναι σπάνιες. Υπάρχουν ε, νομικά κείμενα που εμπνέονται από την Σαρία, αλλά είναι πολύ σπάνιο και βασικά αποτελούν, περιλαμβάνουν τα δικαιώματα ε, κρίσης του δικαστή. Για τη θανατική ποινή μίλησα. Πάλι για τις γυναίκες. Η γυναίκα στη Σαουδική Αραβία παίζει σε ορισμένες περιπτώσεις ηγετικό ρόλο στην ιεραρχία του κράτους. Σήμερα, στο Κοινοβούλιο της Σαουδικής Αραβίας, οι γυναίκες αποτελούν το 20% του Κοινοβουλίου. Σε πολλά ευρωπαϊκά κοινοβούλια ε, οι γυναίκες δεν έφτασαν ποτέ σε αυτό το ποσοστό. Σπάνια βρίσκεις τόσο σημαντική εκπροσώπηση της γυναίκας σε Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Η γυναίκα επίσης μετέχει στις δημοτικές εκλογές μπορεί να γίνει δικηγόρος, μπορεί να ζητήσει την προστασία της από τη δικαιοσύνη لإيماننا بأهمية دور المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية جرى الاهتمام Είμαστε αποφασιστικά πεπισμένοι ότι η γυναίκα παίζει σημαντικό ρόλο στην Σαουδαραβική κοινωνία. Γι' αυτό και δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέμα της γυναίκας. Ίσως στο παρελθόν αυτό να μην συνέβαινε. Σήμερα ωστόσο είμαστε πεπισμένοι για τη χρησιμότητα της βράσης των γυναικών για να έχουμε μια μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα. Τώρα, Twitter, Facebook κλπ. Τα στατιστικά που έχω δείχνουν ότι η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα που χρησιμοποιεί στη χρησιμοποίηση του Twitter. Μόλις τώρα με ρώτησαν και κάτι στο Twitter. Και μας ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό. Ε? Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν υπάρχουν άλλες, ε, είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, ε, λέει ο πρόεδρος, έχουμε τρεις συναδέλφους που θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Ο κύριος Άτκινς από τους ε, ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Καλησπέρα Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι Βρετανός συντηρητικός ευρωβουλευτής και όπως θα ξέρετε η χώρα σας ε, ε, είναι με τη δική μου, είναι, έχουν πάρα πολύ στενούς φιλικούς δεσμούς και έτσι μεταξύ φίλων μπορεί να είμαστε ειλικρινεί. Αν δεν είμαστε ειλικρινεί, τι νόημα έχει φιλία. Έχω τρία ερωτήματα μαζί με άλλους συναδέλφους από όλα τα πολιτικά ε, κόμματα εκφράζω και εγώ τις επιφυλάξει μου για τα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά το, το βρίσκω πραγματικά απίστευτο ότι είναι μόνη χώρα στον κόσμο που οι γυναίκες δεν μπορούν να οδηγούν αυτοκίνητο δημοσίως. Σα το ευχόμουν αυτό για τη γυναίκα μου, αλλά τέλος πάντων. Τώρα η έλλειψη δικαστικής, ε, θρησκευτικής ελευθερίας έχει σχέση με την τήρηση του θρησκευτικού νόμου της Σαρία και όχι τόσο πολύ με ε, την εφαρμογή διοικητικών κανόνων. Είναι σωστό αυτό ή όχι. Δεύτερον, ποια είναι η θέση σας... Ε, What legal and judicial... Ε, ως προς ε, αλλοδαπούς φιλοξενούμενους στη χώρα σας ή ε, οι πολίτες οι οποίοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Εκεί τι γίνεται με την εφαρμογή ή όχι της Σαρία. Και τέλος θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις ανησυχίες μου για τον Μπαχρέιν. Ε, ε, ενδιαφέρουμε ιδιαίτερα για τη θέση, τις αραβικές θέσεις στη Μέση Ανατολή και από ό,τι φαίνεται ε, θα μπορούσε η κατάσταση στο Μπαχρέι να βελτιωθεί, διότι αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι ακολουθεί τη, σωστό, τη σωστή οδό. Ο κύριος Σβένσον από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις, όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι κανένας δεν θα ε, είναι σήμα διακρίσεων ε, και, και μάλιστα θρησκευτικών. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, τη Σουηδία, όπου πολλές, ε, πολλά τζαμιά έχουν χτιστεί και χτίζονται ακόμα. Θα ήταν δυνατόν για χριστιανούς να χτίσουν μια εκκλησία στη Σαουδική Αραβία και πιστεύετε ότι πράγματι δεν υπάρχουν, δεν γίνονται διακρίσεις εναντίον αλόφρισκων όταν το γεγονός είναι κύριε Υπουργέ ότι δεν μπορεί κανείς να εκφράσει ελεύθερα την πίστη του στη Σαουδική Αραβία. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα δεν είναι δυνατόν αυτό να συνάδει ε, με τις διατάξεις του συντάγματος, διότι σύμφωνα με τις συμφωνίες του ΟΗΕ ο καταστατικός χάρτης ορίζει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να, ε, να πιστεύει και να ε, εξασκεί τη θρησκεία του. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ο κύριος Βάγκελ από την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω να, να συγχαρώ τον Υπουργό που ήρθε εδώ στη συνάντησή μας. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία αυτή να ανταλλάξουμε απόψεις. Και είναι πραγματικά σπάνια η ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για τη Σεωδική Αραβία γνωρίζοντας ε, τη σημασία αυτής της χώρας στην περιοχή και στην ε, διεθνή ε, πολιτική σκηνή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που μας απασχολούν δεν απαντήσατε σε ένα ερώτημα που τέθηκε και θα ήθελα να μου, να το θέσω εκ νέου. Κυκλοφορούν φήμες, αλλά όχι μόνο φήμες, ότι πολλοί οπαδοί ε, ακραίων οργανώσεων, όπως αλκαΐδα ε, υποστηρίζονται από διάφορες πηγές ε, της Σαουδικής Αραβίας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτές ε, τις ε, φήμες, τα σχόλια που ακούγονται και θα ήθελα να ξέρω εάν ε, έχετε κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό. Επίσης για τις οργανώσεις των πολιτών, τις αστικές οργανώσεις. Σημείωσα αυτά που είπατε για τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας είναι γεγονός ότι αυτά τα μέσα επικοινωνίας συνήθως ε, χρησιμοποιούνται από νέους, από τη νέα γενιά και οργανώσεις πολιτών. Έχετε πολύ περιοριστική νομοθεσία όσον αφορά τη χρήση τους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η νομοθεσία δημιουργεί πολλά προβλήματα στην, ε, στους πολίτες και στην κοινωνία. Ε, και δεν συνάδει αυτό με την ελευθερία έκφρασης. Ε, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο, βλέπετε να υπάρχει κάποιο περιθώριο φιλελευθεροποίησης αυτών των μέσων. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. آتي في Καταρχάς, για την πρώτη ερώτηση, τα δικαιώματα των γυναικών. Σας εκπλήσει το ότι δεν οδηγούν αυτοκίνητα γυναίκες στην Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει κανένα γενικό νομοθετικό ή συνταγματικό κείμενο ή κανονισμός που απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγούν στη Σαουδική Αραβία. Πιστεύω ότι η συνταγματικο κειμενο η κανονισμο που απαγορευει στις γυναικες να οδηγουν στη σαουδικη αραβια πιστευω οτι η γυναικα δεν οδηγεί, απέχει από τον οδηγήσει γιατί δεν το θέλει. Είναι ένα μοντέλο που σχετίζεται με την κουλτούρα της κοινωνίας η γυναίκα είναι που δέχεται, η γυναίκα είναι που ε, δεν δέχεται να οδηγήσει. Έτσι είναι φτιαγμένη η κοινωνία μας, έτσι εξελίχθηκε. Δεν υπάρχει ωστόσο νομικό κείμενο που να απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγήσουν. Ούτε υπάρχει κείμενο που να επιβάλλει στις γυναίκες να οδηγούν. Εάν λοιπόν η γυναίκα σήμερα οι περισσότερες γυναίκες σε Σαουδική Αραβία πούν αύριο θέλουμε να οδηγήσουν, δεν θα πει κανείς όχι. Επιβεβαιώνω, δεν υπάρχει απαγόρευση στο σύνταγμα, στο κανονικό δίκαιο της Σαουδικής Αραβίας οπουδήποτε αλλού που να απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγήσουν. Απλά η παράδοση είναι. Η γυναίκα το θέλησε. Να, η γυναίκα θέλει να μην οδηγεί. Για τη δεύτερη ερώτηση, τους περιορισμούς στην ε, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εγώ επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, διάφανη, Κανείς δεν έχει την υποχρέωση να... Την, κανείς δεν αποφεύγει, δεν μπορεί να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν χωριστές ελεύθερες διαδικασίες ποινικού χαρακτήρα, αστικού χαρακτήρα, δημόσιες ε, συνεδριάσεις πάντα, παρουσία των δημοσιογράφων των μέσων, όλοι έχουν πρόσβαση και μπορούν να το μεταφέρουν σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Ο καθένας μπορεί να μετάσχει στην διαδικασία ή να πάει σε, κάποια σε κάποιο δικαστήριο να παρακολουθήσει την δικαιοσύνη. Αυτό είναι βασική αρχή. Η δημοσιότητα και οι ανοιχτές διαδικασίες είναι βάση της διαδικασίας μας. Επιβεβαιώνω επίσης ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση στα δικαστήρια μεταξύ Σαουδαράβων και μη, μουσουλμάνων και μη. Ένα από τα θεμέλια της δικαιοσύνης είναι μη διάκριση. Δικαιοσύνη για όλους χωρίς καμία διάκριση. Αν έχετε συγκεκριμένο παράδειγμα, εδώ ή αλλού, που δείχνει ότι υπάρχουν διακρίσεις, θα ήμουν έτοιμος να το δω μαζί σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακούτε ε, ότι στηρίζεστε σε στερεότυπα, σε προκαταλήψεις Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συγκεκριμένη που ε, διαφοροποιεί αυτό που σας είπα. Ολόκληρο το νομικό μας οπλοστάσιο επιβεβαιώνει την αλήθεια αυτών που σας έχω πει. Φέρετε μου ένα παράδειγμα, να σας πω, να το δω και να σας πω. Ναι, έκανα λάθος, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα για το Μπαχρέιν. Μπορεί να ρωτήσετε και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μου. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια αμυντική συμφωνία μεταξύ των χωρών συνεργασίας του κόλπου, του Περσικού κόλπου. Και ορισμένες από τις ε, διατάξεις αυτές αναπερίπτωση τις εφαρμόζουμε εφόσον δεν αντιβαίνουν στις συνταγματικές αρχές ε, κάθε χώρας. Είτε πρόκειται για χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, είτε για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες. Τώρα για τις θρησκευτικέ πρακτικές της Σαουδική Αραβία. Ο κόσμος σήμερα έχει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους στον πλανήτη. Η μεγάλη πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τις εκθέσεις, τις στατιστικές και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και του σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία τους, επαναλαμβάνω, θεωρούν ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία γη, μία χώρα με αποκλειστικό σημείο αναφορά στην ε, λατρεία του Ισλάμ. Η με, πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων στην γη θεωρούν ότι η Σαουδική Αραβία, είναι μια χώρα που, που, έχει είναι αποκλειστικά ε, προσανατολισμένη στην λατρεία του Ισλάμ. Και ρωτώ, το Βατικανό θα δεχόταν να έρθει ένας μουσουλμάνος να χτίσει μία, ένα τζαμί εκεί. Πρόκειται για μία ειδική κατάσταση μια ειδική περιοχής του κόσμου. Ωστόσο, κανείς δεν εμποδίζεται να ασκήσει την θρησκευτική του λατρεία στη γη μας. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να υπάρξουν κτίρια μη μουσουλμανικά στην γη μας. Αυτό ε, δεν συμβαίνει αλλού. Οι υπόλοιπες, ε, στις υπόλοιπες ε, Ισλαμικές χώρες ε, με την εξαίρεση της Σαουδικής Αραβίας υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής εκκλησιών. Εμείς θεωρούμε ότι η Σαουδική Αραβία, ο χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι ένας χώρος αποκλειστικής ε, λατρείας του Ισλάμ. Σας παρακαλώ να το δεχτείτε αυτό, να καταλάβετε αυτή την διάσταση. Έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε τη γη αυτή μόνο για, την λατρεία του, για τη μουσουλμανική λατρεία και παρακαλούμε, ζητάμε να το σεβαστείτε. Πρόκειται για έναν χώρο που είναι ιερός για 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Στις υπόλοιπες ε, οι μουσουλμανικές χώρες δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την κατασκευή ε, χώρων λατρείας άλλων θρησκευμάτων. Ξέχασα να απαντήσω σε μία ερώτηση. της φήμες για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή ακραίων ε, οργανώσεων στον κόσμο. Εδώ και δέκα χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε κατά της τρομοκρατίας στη Σαουδική Αραβία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα στον κόσμο που έχει υποφέρει περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία. Τι μας λέτε λοιπόν ότι χρηματοδοτούμε το Αυτούς που μας βλάπτουν θα χρηματοδοτήσουμε. Να σας πω ότι στην Σαουδική Αραβία υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν τη χρηματοδότηση αλλοδαπών οργανώσεων. Ο νόμος απαγορεύει την χρηματοδότηση αλλοδαπής οργάνωσης χωρίς άδεια. Εγώ ο ίδιος εξέτασα αποφάσεις κατά ατόμων που ξεπέρασαν το όριό τους και χρηματοδοτούν αλλοδαπές δραστηριότητες. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι υπεύθυνη για τέτοιες ε, ε, συμπεριφορές. Και όποιος το κάνει οδηγείται στη δικαιοσύνη. Νομίζω επίσης ότι υπάρχουν χώρες στον κόσμο που υιοθετούν νόμους για να χτυπήσουν την τρομοκρατία. Οι χώρες αυτές, μπορώ να σας πω, ότι έκαναν λιγότερο από αυτά που κάναμε εμείς στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Η βούλησή μας κατά της τρομοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν θα καμφθούμε στη μάχη κατά της δημοκρατίας τόσο εντός όσο και εκτός. Να σας επιβεβαιώσω επίσης το ίδιο θέμα ότι εμείς καταβάλαμε πάρα πολλές προσπάθειες και εξελιχθήκαμε σημαντικά σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίησή μας για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών. Κάναμε πολλά για την κοινωνία των πολιτών. Τίποτα στη Σαουδική Αραβία δεν εμποδίζει την εφαρμογή, τη λειτουργία φιλανθρωπικών οργανώσεων οργανώσεων που έχουν ε, μη κερδοσκοπικό κοινωνικό χαρακτήρα, τη λειτουργία συνδικάτων. Υπάρχουν οργανώσεις δικαιωμάτων ανθρώπου με πολύ στενούς δεσμούς με άλλες ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ εξοχότατε για τις, απα... για σας. Πολύ σύντομα ο κύριος Πέτερη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνη, ε, ζητώ συγγνώμη που μόλις ήρθα στην ε, αίθουσα. Αλλά όσον αφορά αυτά που είπατε για την ανεξιθρησκεία, θα ήθελα κάτι να προσθέσω. Είπατε ότι στο Βατι... και στο Βατικανό δεν χτίζεται τζαμί. Αυτό σημαίνει ότι εσείς ε, θεωρείτε ολόκληρη τη Σαουδική Αραβία ως ε, μουσουλμανικό Βατικανό. Εάν στη Μέκα και στη Μεντίνα δεν έχετε χριστιανικές εκκλησίες, το κατανοώ απολύτως. Αλλά όλη η επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας και το να δηλώνεται ότι δεν μπορεί να χτιστεί ποθενά εκκλησία, το θεωρώ απαράδεκτο. Δεύτερον, Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει ακόμα ένας νόμος στη Σαουδική Αραβία που λέει όταν ένας μουσουλμάνος αλλάξει θρησκεία και θέλει ας πούμε να σπαστεί μια άλλη θρησκεία, το χριστιανισμό. Ε, γι' αυτό το αδί, είναι αδίκημα που επιφέρει τη θανατική ποινή. هل الفلسفة في المنع هي فلسفة مساحة أو فلسفة مبدأ؟ هل منع إقامة مساجد أو جوامع في الفاتيكان هي مساحة أو فلسفة مبدأ؟ φιλοσοφία μας σχετίζεται ε, το ερώτημα που σας θέτω είναι η φιλοσοφία που έχουμε για την απαγόρευση κατασκευής ε, ε τόπων λατρείας ε, στηρίζεται στο Βατικανό στηρίζεται μόνο στο, στην έκταση ή και σε θέματα αρχής γιατί αν είναι μόνο στην έκταση είναι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω ότι η απαγόρευση είναι επί της αρχής, δηλαδή απαγορεύεται η κατασκευή τόπων λατρείας σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο που είναι αφιερωμένο σε κάτι το ειδικό και που δεν μπορεί να δεχθεί άλλες χρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να πειράξουμε την συνείδηση 1,5 εκατομμυρίου ε, μουσουλμάνων. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά πρόκειται για μία φιλοσοφία, για, μία, για ένα αξίωμα ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία γη αποκριστική για μία συγκεκριμένη λατρεία, μία γη που επελέγει για να ε, φιλοξενήσει τα ιερά ε, τεμένη των ε, ε, μουσουλμάνων. Και δεν είναι θέμα έκτασης, αλλά θέμα αρχής για την ε, θανατική καταδίκη των αποστατών. Στο Ισλάμ ο αποστάτης καταδικάζεται σε θάνατο ή μη μόνο αν προβεί σε εσχάτη προδοσία των ε, ιερών θέσεων του Ισλάμ. Η εσχάτη προδοσία στη Σαουδική Αραβία αλλά και αλλού τιμωρείται με το θάνατο. Σε εμά ωστόσο θανατική απόφαση κατά κάποιου που χαρακτηρίζεται ως αποστάτης απονέμεται μόνο με, για εσχάτη προδοσία και μετά από διεξοδική εξέταση. Πείτε μου, έχετε παραδείγματα συγκεκριμένες περιπτώσεις αποστατών είτε Σαουδαραβών είτε μη που καταδικάστηκαν με θανατική ποινή. Γράψτε μου, πείτε μου, δώστε μου συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όχι άκουσα, είπα, μου παν. Μιλάμε για νομικές αρχές. Μιλώ για δικαιοσύνη. πρέπει να ερευνήσουμε, να εξετάσουμε, να βρούμε. Δεν ε, πρέπει να στηρίζεστε μόνο σε φήμες. για να κρίνετε με τόσο σοβαρό τρόπο. οι περιπτώσεις εξετάζονται προσεκτικά. Και αν στη Σαουδική Αραβία υπάρξουν εσφαλμένες κακές πρακτικές, δεν θα τις ανοιχτώ. Αλλά να αποδειχτεί πρώτα. Γνωρίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια. Γι' αυτό και αλλάζουν οι νόμοι. Γι' αυτό γίνονται δημοψηφίσματα για συντάγματα. Κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει την απόλυτη, την απόλυτη αλήθεια. Σας ευχαριστούμε. Εξοχότατε. Νομίζω ότι ήταν καρποφόρα η ευκαιρία αυτή και για τις δύο πλευρές να γνωρίσουν οι μεν τον τρόπο σκέψης των δε και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Εξοχότατε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen. Ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, καθίστε. Wir wollen kurz... Να σας ενημερώσουμε με λίγα λόγια για την διακυβουνοβουλευτική διάσκεψη CFSP και CSTP στο Δουβλίνο Είναι παρόν και ο Πατ Μπριν που είναι πρόεδρος της ε, Ιρλανδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα ασφάλειας και εξωτερικών κτλ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, καθώς επίσης ευχαριστώ και για την διάσκεψη, καθώς και για την θαυμάσια φιλοξενία που μας προσέφεραν στη διάρκεια της διασκέψεως, η οποία και από άποψη ουσιώδου περιεχόμενου αλλά και από την άποψη προσωπικών επαφών. Ήταν θαυμάσια ευκαιρία και γνωρίζω βεβαίως τι δουλειά σημαίνει μια τέτοια εκδήλωση. Ακόμα και αν κάποιο έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι δεν γνωρίζει αυτομάτω πώ ε, λειτουργεί και πώ σκέπτεται η Ιρλανδία. Η διάσκεψη αυτή λοιπόν έγινε για δεύτερη φορά στις 25-26 Μαρτίου στο Δουβλίνο, αμέσως μετά από την συνάντηση του Γκίμνιχ. Ήταν παρούσα και η Αντιπρόεδρος Άστον, καθώς και ο Ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και ο Ιρλανδός Υπουργός Άμυνας, καθώς και αξιωματούχοι και επιστήμονες και ο κ. Σκοπόφσκι της ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Για πρώτη φορά ε, χωρίστηκε η εργασία σε δύο ομάδες εργασίας. Ήταν σημαντικό αυτό γιατί έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους συναδέλφους του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων δόθηκε η ευκαιρία και ο χρόνος να εγκύψουν εντατικότερα σε επιμέρους θέματα από ό,τι θα ήταν δυνατό σε μεγάλες ε, συζητήσεις ε, στην Ολομέλεια της διασκέψεως. Μιλήσαμε για το κέρας της Αφρικής, για την σύγκρουση στην Εγγύς Ανατολή. Αυτά συζητήθηκαν και στις δύο ομάδες εργασίας. Ο κ. Ντονζόν ήταν ε, εισηγητής για, την, για το πρώτο αυτό εργαστήριο και είναι καλό στη βάση της ιδέας αυτής που εφάρμοσαν οι Ιρλανδοί συνάδελφοί μας Νομίζω ότι αυτή η ιδέα λοιπόν είναι καλό να συνεχιστεί. Και από όσο γνωρίζω η Λιθουανική Προεδρία έχει την πρόθεση να υιοθετήσει το μοντέλο του Δουβλίνου και για την διάσκεψη που θα διεξαχθεί τον επόμενο Σεπτέμβρη. συμφωνήσαμε να εξετάσουμε και πάλι με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η διάσκεψη. Υποβλήθηκαν κάποιε πρώτε ιδέε και δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασία που θα αρχίσει τι εργασίε τη υπό την αιγίδα τη Ιρλανδική Προεδρία και η ομάδα εργασία αυτή αποτελείται από Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα την Τρόικα συν, αν μπορώ να το πω έτσι, Τρόικα συν. Οι Κύπροι είναι μέσα διότι αυτοί άρχισαν και με τους Ιταλούς θα ολοκληρώσουμε. Ήταν σωστό λοιπόν να έχουμε όλη αυτή την ομάδα ώστε να μπορούν να γίνουν προτάσεις για το πώς θα εξελιχθεί η διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Εμείς του Ευρωκοινοβουλίου τονίσαμε ότι αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας των Προέδρων Κοινοβουλίων στην Βαρσοβία. Δεν χρειάζεται να επανεπινοήσουμε ε, την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Ορισμένε βασικέ αρχέ μπορούν να παραμείνουν. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου οι Κύπροι φίλοι μας αρχικά είχαν προωθήσει μια ιδέα. Είχαν προτείνει δηλαδή να κάνουμε μια fact-finding mission, μια εξεταστική των πραγμάτων αποστολή για θέματα γειτονικής πολιτικής, πολιτικής γειτονίας της Μεσογείου. Αν αρχίσουμε έτσι όμως, αν κάθε χώρα προτείνει και γίνεται μια εξεταστική των πραγμάτων αποστολή, τότε η διακοινοβουλευτική διάσκεψη θα καταλήξει στην εγγραφή ταξιδιών κάτι το οποίο θα υπερεπιβαρύνει τη διοίκηση και της χώρας αυτής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Κάθε βέβαια Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να οργανώσει τέτοια αποστολή και να προσκαλέσει και προσώπους άλλων κοινοβουλίων. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να συζητηθεί χωρίς όμως να φτιάξουμε ένα ειδικό μηχανισμό για τέτοιες αποστολές, ένα ταξιδιωτικό μηχανισμό εντός εισαγωγικών. Την έκθεση θα την υποβάλουμε και στον πρόεδρο Σούλτς με την υπόδειξη ότι θα πρέπει την διεύθυνση να αναλαμβάνει στο μέλλον η Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσει. Παρανοήσει που υπήρξαν και στι ορισμένε χώρες μέλη που θεώρησαν ότι είναι μια συνέχεια της παλιάς Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δεν, σημαίνει, δεν συμβαίνει αυτό. Πρόκειται για διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Η επόμενη λοιπόν ε, διάσκεψη θα γίνει 4 6 ενάτου στην Βίλνιους. Θα συμμετάσχουν στη 16 μελή σύνθεση οι πολιτικές ομάδες κατά τη γνωστή κατανομή. Στο Δουβλίνο ήταν 15 παρόντες και θα παρακαλέσω τις χώρες μέλη, τι, συγγνώμη, θα παρακαλέσω τις πολιτικές ομάδες από τώρα να εγκύψουν στο θέμα. Γιατί 4 6 Σεπτεμβρίου είναι αμέσως μετά τις θερινέ διακοπέ. Άρα πρέπει από τώρα να οριστούν τα μέλη, ώστε να είναι προετοιμασμένη καλά η διάσκεψη. Εγώ θα χαρώ πάντω εάν ο Πατ Μπριν θελήσει να κάνει και αυτός λίγες παρατηρήσεις για την ε, διάσκεψη και εκφράζω και πάλι τις ευχαριστίες μου για τη θαυμάσια συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ περιμένω με υπομονησία την, ε, το συνέδριο στο Βίλνιου, που πολύ σωστά είπατε θα πραγματοποιηθεί αμέσω μετά τις θερινές διακοπές. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια σε σχέση με το πρόσφατο συνέδριο του Δουβλίνου. Πράγματι, Πήρα πολλά email μετά το συνέδριο και από αυτά συνάγω το συμπέρασμα ότι πήγε πολύ καλά το συνέδριο. Βέβαια, είμαστε στην αναπτυξιακή φάση. Το πρώτο συνέδριο έγινε στην Κύπρο, στην Πάφο, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και αυτή η διάσκεψη ουσιαστικά είναι η πρώτη του είδους της με 230 συμμετέχοντες. Ήταν πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, για όλους μας ε, στο Δουβλίνο ουσιαστικά να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που επιτελέστηκε ήδη στην Κύπρο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή εθνικών βουλευτών αλλά και ευρωβουλευτών ήταν και πάλι σημαντικό για μας και χρειαζόμαστε τους βουλευτές αυτούς ε, στο συνέδριο, στην διάσκεψη αυτή και έπρεπε να έχουν λόγο γιατί περί αυτού πρόκειται σε τέτοιες διασκέψεις. Επίσης θελήσαμε να ε, οργανώσουμε κάποια εργαστήρια που όπως είπατε και εσείς πέτυχαν πολύ. Ε, οι εργασίες τους ήταν πολύ επιτυχημένες. Διαλέξαμε θέματα που ενδιέφεραν τους βουλευτές και ήταν βέβαια στήματα της επικαιρότητα, διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Δόθηκε τεράστια έμφαση στη Συρία και στην αναπτυξιακή βοήθεια που νομίζω και αυτό ήταν ένα σημαντικό σκέλος. Σημαντικά λοιπόν τα θέματα, ακολουθήσαμε μια γενική προσέγγιση και για το Μεσανατολικό και νομίζω ότι και ο κύριος Άντες Ράιν και είχε μια πολύ σημαντική συμβολή ε, στις συνεδριάσεις και στα εργαστήρια. Σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά εργαστήρια τώρα, κύριε Πρόεδρε, νομίζω είπατε και εσείς ότι η λιθουανική κυβέρνηση υιοθετεί το μοντέλο αυτό, είναι σημαντικό από τη στιγμή που ε, συνεδριάζουν από κοινού τόσοι πολλοί βουλευτέ, καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα διαλύματα και στο πλαίσιο εργαστηρίου να συζητούνται οι ειδικέ, οι ιδιαίτερε ανάγκε. Αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σωστά επίση είπατε ότι είχαμε και αυτή την ad hoc επιτροπή, την ειδική επιτροπή που ε, θα δει πώ λειτουργήσε η όλη διάσκεψη. Θα γίνει αυτή η αναθεώρηση στη Ρώμη σε δύο χρόνια, όπω πολύ σωστά είπατε και εσεί. Και αυτή η ad hoc επιτροπή θα δει τι γίνεται ε, στις διασκέψεις ε, που διοργανώθηκαν μέσα στα τελευταία δυόμιση χρόνια για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πεπραγμένα και να έχουν και επαναλαμβάνω λόγο οι βουλευτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινέστατα για τις πολύ γενικέ παρατηρήσεις σας. Ε, ο Νταν Νέβολες που είναι μέλος Επιτροπής Εξωτερικών και εγώ βλέπουμε πάρα πολύ με πολύ ενδιαφέρον και από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του δικού σας ε, κοινοβουλίου. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ήμασταν εδώ. Και βέβαια προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μελλοντικό μας έργο και περιμένουμε επίσης με υπομονησία να βοηθήσουμε και τους λιθανούς συναδέλφους μας και γενικώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της διάσκεψης της Λιθουανία το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας καθώς και για την συνεργασία, όπως είπα και πριν. Ξέχασα να πω ποιο θα είναι το κύριο θέμα της διασκέψεως του Σεπτεμβρίου. Θα είναι η αμυντική, αμυντική πολιτική και πολιτική εξωτερικών για την διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Και κύριε Ντανζόν θα έχουμε και τη στενή συνεργασία γι' αυτό έτσι ώστε να καταλήξουμε εκεί να προβάλλουμε τις απόψεις μας με συνεκτικό τρόπο. Τώρα, υπάρχουν παρακαλώ σχόλια ή παρατηρήσεις. Ορίστε εσείς κύριε παρακαλώ. Δεν περίμενα ότι θα ήμουν ο μόνος που θα ήθελα να σχολιάσει, αλλά νιώθω ιδιαίτερα προνομιούχος που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε και με επιλέξατε. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ άκρος ηρωνικό το γεγονός ε, αυτό, αυτή η διάσκεψη για την ΚΕΠΑ να συνεδρίασε για τελευταία φορά στην Κύπρο. Στο Δουβλίνο προσφάτως και επόμενη συνεδρίαση στη Ρώμη. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος, στο Βίλνιους. Η Ρώμη πού, πού μπήκε. Α, σε δύο χρόνια, μάλιστα. Πρόεδρος, ναι, μετά τις εκλογές. Δεν θα έχετε πρόβλημα, μπορείτε να πάτε. Α, μάλιστα. Ωραία, τα μπέρδεψα. Λοιπόν, στη Ρώμη είναι μεθεπόμενη. Αυτό που άκουσα στην παρουσίαση ε, Κύπρος, Δουβλίνο, Ρώμη. Για σκεφτείτε, τρεις χώρες. Υπάρχουν τρεις χώρες που να έχουν καταστραφεί περισσότερο από αυτή την... Ε, καταστροφική μηχανή ε, της οικονομικής κρίσης παραπάνω από αυτές τις τρεις ε, χώρες. Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία που διοργανώθηκαν αυτές ε, οι συνεδριάσεις εκεί. Πραγματικά με ξεπερνάει και εμένα. Ε, δηλαδή είναι πιο σατερικό δεν γίνεται, πιο τραγική ηρωνία δεν γίνεται. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Βλέποντας ε, την πρόταση που έχω μπροστά μου, το σχέδιο έκθεσης, αν περί αυτού πρόκειται, ως πρόεδρος είπατε ότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και μέσα είναι το βασικό θέμα. Το βλέπουμε εδώ. Λέτε εδώ στήριξη πολιτική ηγεσία ε, στον τομέα της ΚΕΠΑ. Στο H και στο I λέτε για μάχη με ομάδες ευρωπαϊκές battle groups. Στο J λέτε να υπάρχουν μόνιμα στρατηγία αρχηγεία στις Βρυξέλλες και μετά τι λέτε στη συνέχεια. Στρατιωτικά μέσα πριν από τις κοινέ στρατηγικές επιλογές της Ένωσης. Ή λέτε στο 17 να δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό αρχηγείο μόνιμο. Και είναι ανησυχητικό. Βέβαια και πάλι και τραγική ηρωνία είναι το ότι συζητάτε για αυτή την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και για έναν επιτετραμένο που θα πρέπει να έχει κάθε προσωπή. Αυτό ο στρατιωτικό ακόλουθο ε, ή επιτετραμένο, τι είναι αυτό το πράγμα. Και όλο το κείμενο, αν το διαβάσει κανεί, βρήθη εκφράσεων ε, που ε, αναφέρονται στην ΚΕΠΑ. Δεν έχετε όμως απολύτως καμία ε, εντολή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χώρα. Όταν υπήρχε στην πρόσφατη ανάφλεξη που είχαμε στη Λιβύη, στην τελευταία εκεί τέλος πάντων, ανάφλεξη. Είχαμε έξι ευρωπαϊκά κράτη τα οποία ήταν σε μια συμμαχία, εκ των οποίων τα δύο δεν ήταν καν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι και εκεί είναι το σημαντικό για μένα. Όταν εσείς και οι συνάδελφοί σας θα προσπαθήσετε να επιδιώξετε τις φεντεραλιστικές σας φαντασίες, φαντασιώσεις και δεν έχετε καμία εντολή γι' αυτό και είναι και αστείο και περίεργο όπως είπα και πριν αλλά ε, είναι και σοβαρό το εξής. Αν αυτή η αδίστακτη πολιτική συνεχιστεί, δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και ένας ευρωπαϊκός στρατός, τελικά το αποτέλεσμα θα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε να φύγουν από το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να μην είναι τότε μία από αυτές η δική μου χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να βασιστεί στα δικά τη αμυντικά μέσα, στη δική τη άμυνα. Ωραία και καλά είναι να προσπαθείτε ίσω και δημοσίε δαπάνε να ικανοποιήσετε αυτέ τι φαντασιώσει σα και να τι πραγματοποιήσετε. Αλλά από αυτή την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα πρέπει να σα πω ότι θα απειληθεί η ευημερία και η ασφάλεια καθενό Ευρωπαίου πολίτη, καθεμίας ευρωπαϊκής χώρας. Είτε ανήκει αυτή στην Ένωση είτε όχι. I suggest, I sir, Robert Atkins. I uh, καλύτερα απαντήσετε στα πολύ σοβαρά επιχειρήματά μου, εάν είστε σε θέση να το κάνετε, που δεν το πιστεύω κιόλας. Οι φαντασιώσεις μου δεν είναι φαντασιώσεις για μάχη με ομάδες, είναι διαφορετικές. Δεύτερο, Εντό τη τρέχουσα εβδομάδα θα σα δώσω ένα αντίγραφο τη συνθήκη τη Λισαβόνα και θα τα βρείτε, του περισσότερου αυτού όρου θα του βρείτε στη συνθήκη τη Λισαβόνα μαζί και τα battle groups. Δεν έχετε το λόγο τώρα. Δεν έχετε το λόγο τώρα. Δεν έχετε το λόγο. Είμαστε ευγενεί και μιλούμε καθένα με τη σειρά του. Battle groups, συντονισμό, στρατιωτικά μέσα, όλα αυτά είναι μέσα στην συνθήκη. Το κέρας Αφρικής, ήταν πολύ καλά αυτά που κάναμε για τη Βρετανική ναυτιλία και το Βρετανικό εμπόριο. Προστατέψαμε τότε το Βρετανικό εμπόριο, γιατί δεν είσαστε πια ανατολικά του Σουέζ, από ό,τι έχω μάθει, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει, δηλαδή εδώ και μερικέ δεκαετίε. Ξαναδιαβάστε λοιπόν λίγο τη συνθήκη, είναι προ το συμφέρον σα. Είναι η συνθήκη τη Αβώνα. Και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων απεφάσισαν να μιλήσουν για τα πράγματα αυτά τον Δεκέμβρη. Και ω κοινοβούλιο λοιπόν τα συζητούμε και εμείς μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ευθύνη και της εθνικής Ευθύνη. Γι' αυτό και έχουμε οργανώσει το όργανο αυτό Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αλληλοενημερωθούμε με κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τις εθνικές διοικήσεις και γραφειοκρατίες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προβλέπεται ως διακοινοβουλευτική διάσκεψη της ESTP από, που έχει αποφασιστεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην συνθήκη της Αφώνας. Θα σας κάνω δώρο ένα αντίγραφο, το οποίο μάλιστα το έχει κυρώσει η Βουλή των Κοινοτήτων στο Westminster. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τα σταματήσετε αυτά. Το δε ΝΑΤΟ είναι επίσημες στη συνθήκη. Είναι πρωτογενές δίκαιο. Έχει αποφασιστεί να γίνει μαζί με τον ΝΑΤΟ. Αν δεν οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να έχουν ισχυρή Ευρώπη, νομίζω ότι ενδιαφέρονται, διότι η ισχυρή Ευρώπη μπορεί να του βοηθήσει. Και εδώ τα κάνουμε αυτά τα πράγματα όχι στρεφόμενοι κατά των Αμερικανών, αλλά ίσω κατά των δικών σα φαντασιώσεων. Ο κ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Πρώτο, πρέπει κανείς να είναι αντικειμενικός. Όταν μιλεί κανείς για φαντασιώσεις, ας μην αντιπαραβάλλετε εσείς τις δικές σας φαντασιώσεις στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι είναι. Είναι η συνθήκη της Λισαβόνας που μιλεί για κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρόκειται λοιπόν για πραγματικότητα ε, και την έχουν κυρώσει οι χώρες μέλη. Δεύτερο, η συνθήκη της Λισαβόνας αναπτύσσοντας αυτή την κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και Άμυνας δεν αμφισβητεί ουδαμός τον ρόλο Ολυκρατικής Συμμαχίας. Σας υπενθυμίζω ότι ένας αριθμός χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ και επιθυμούν και αυτές να μπουν σε μια ε, αρχιτεκτονική συμμαχία. Τρίτο και πιο σημαντικό από τις φαντασιώσεις σας, ήδη σήμερα και εδώ και τρία χρόνια η Μεγάλη Βρετανία υποδέχεται στο έδαφος της λειτουργικό επιτελείο επικεφαλής του οποίου είναι Βρετανός Ναύαρχος και κανείς δεν έχει αντιταχθεί στις αποστολές της ε, κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυλας για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ανοιχτά της Ομαλίας και έξω από τον κόλπο του Άντεν. Και εσείς ε, θέλετε να απαντήσετε στον κόμιτα του Ντάγμορ, κύριε Πέτερινγκ κάθε παρατήρηση εγώ την λαμβάνω σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό θα πω στο συναδελφό μου Dartmouth. Ο ισχυρότερος συνήγορος της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας και του, Αμερικανικού, και του Ευρωπαϊκού στρατού ήταν ο Τζον Φώστερ Ντάλλες, προς εξωτερικών των ΗΠΑ τη δεκαετία του 50. Πρώτο. Το δεύτερο, αγαπητέ φίλε, έχω μεγάλη συμπάθεια για, την, ε, για το Ενωμένο Βασίλειο και γι' αυτό επιθυμώ το Ενωμένο Βασίλειο να παραμείνει ένα ενιαίο σύνολο και να μην αποσχιστούν τμήματά του. Σας υπενθυμίζω όμως, όταν δείχνετε την αποστροφή σας προς την Ευρώπη και, την, και τις Βρυξέλλες, ίσως να συμβάλλετε έτσι στο να αποχαιρετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο η Σκοτία μέσω δημοψηφίσματος, ο Ρόμπερτ. Εγώ δεν θεωρώ ότι θέλω να συμμετάσχω στην κοινή άμυνα και ασφάλεια, ούτε μου αρέσουν όμω αυτά που είπε ο συνάδελφό μου από το κόμμα ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεργασία, όπου μπορεί να γίνει αυτή, σε κάθε επίπεδο είναι καλοδεχόμενη. Ένα από του συναδέλφου μου είπε προηγουμένω, μάλιστα εσεί ο ίδιο κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα τη πειρατεία στο κέρα τη Αφρική και σε άλλε κοντινέ περιοχέ που μεγάλο ζημίωσαν το βρετανικό εμπόριο. Εφόσον θέλουμε να συζητήσουμε, ας τα κάνουμε τα πράγματα αυτά, ας τα πούμε τα πράγματα αυτά ψύχρεμα και αντικειμενικά. Και ας μην επιτρέψουμε να ξεφύγουν κάποιοι λόγω προκαταλήψεων. Ο ταξιάρχος Τζέφι Βαν Όρντεν ήταν στην CDSP για πολλά χρόνια και ε, ήταν αντίπαλος, συγγνώμη, αντίπαλος της ε, CDSP για πολλά χρόνια, αλλά τα έκανε με πολιτισμένο τρόπο να έρχεται τώρα ένα μέλος της Βουλής των Λόρδων δεν είναι τρόπος να μιλεί έτσι. Ορίστε κύριε Κόμη. Ε, ευχαριστώ για την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε. Εγώ ανέφερα 20 περίπου παραθέσεις από το σχέδιο εκθέσεως και όσα είπα στηρίζονται στα γεγονότα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Πρόκειται να εξοπλιστεί με στρατιωτικά μέσα και εφιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσοχή της Επιτροπής σας στο γεγονός αυτό. Δεν είχα κανένα, ε, καμία απολύτως πρόθεση ε, να ε, κάνω φασαρία. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα λέει αυτά η έκθεση. Είπα όμως ότι τα λέει, καλά κάνει και τα λέει η έκθεση. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Για το θέμα της μεσής διδάξης υπαρχών 5. Ήδη η κυρία Λούνατσεκ αρχίζει και με αγρίο κοιτάζει. Ε, καλή επιτυχία στο έργο σας, Πατ, και στην ομάδα σας. Όμως πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλα μέλη να ομιλήσουν. Θα σας δώσω το λόγο όμως να κάνετε την εισαγωγή πριν να χρειαστεί να φύγετε. Ακούστε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Αρχικά η ΑΕΔ ήταν στην ημερήσια διάταξη, προβλεπόταν όμως για τις 4 και άλλαξε αυτό ε, τελευταία. Εγώ όμως έπρεπε να αντικαθιστώ την ε, Φραντσίσκα Μπνάτνερ ε, για ε, την ΑΕΔ και στις 5 προεδρεύω μια άλλη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε λοιπόν το λόγο για να σας θέσω όλα αυτά τα ζητήματα πολύ πολύ γρήγορα. Συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις συζητητές, συζητήσαμε τις συμβαστικές προτάσεις, υπάρχουν ακόμη κάποια εκκρεμή θέματα και θα σας πω ότι είναι σημαντικό για για μας και για την ομάδα μας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή. Η έκθεση έχει προχωρήσει. Είχαμε ε, ακούσει κάποιες κριτικές για την ΕΙΕΔ αλλά έχουμε επικροτήσει και το έργο της Κάθρι Άστον μέχρι τώρα που δεν ήταν εύκολη δουλειά τη. Ωστόσο, η έκθεση αυτή πολύ ξεκάθαρα δείχνει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μεταρρυθμιστεί η ΑΕΔ για διάφορα, σε διάφορου τομεί. και στου συμβιβασμού ε, νομίζω ότι Έχουμε κάνει καλές προτάσεις για τα βασικά θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ε, συμβαστική τροπολογία, την υπαριθμόν 7, όπου η Φραντσίσκα Μπραντνερ μου ζήτησε, και το έχω ελέγξει με τον κύριο Γκουαλτιέρη, που γίνεται λόγος για την ανάπτυξη περαιτέρω και κατάλληλης δομής που θα περιλαμβάνει και το σκέλος της πρόληψης συγκρούσεων. Η κυρία Μπράτνερ Λέει να το πούμε κάπως σαν ε, διεύθυνση διαχείρισης κρίσεων. Εσείς είπατε να είναι συμβούλιο, ε, board ή directorate. Για να το πούμε ε, διεύθυνση, ουσιαστικά θέλουμε να προωθήσουμε την συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ ομάδων. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείτε να το εξετάσετε και να το λάβετε ενδεχομένω υπόψη. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι εκφράζει κάτι διαφορετικό ως ιδέα σε σχέση με την αρχική πρόταση. Για τα άλλα σημεία θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις τροπολογίες για τις οποίες ελπίζω να μας στηρίξουν οι εισηγητές αλλά και άλλοι συνάδελφοι από την Επιτροπή εδώ αύριο. Μία τροπολογία η 134 ε, αναφέρεται στην μεγαλύτερη ευελιξία Μιλάει για αναθεώρηση των κανόνων για τις αποφάσεις, για τον προγραμματισμό και τις δαπάνες για τα μέσα εξωτερικής βοήθειας και αυτό είναι σημαντικό για το παρελθόν μας δημιούργησε κάποια προβλήματα, ακριβώς αυτή η έλλειψη ευελιξίας ε, στην εξωτερική βοήθεια και στα χρηματοδοτικά μέσα. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να μας στηρίξουν. Επίσης, όπως αναφέρθηκε η προηγούμενη συζήτηση, Έχουμε αυτούς τους ακόλουθους ή επιτετραμένους ασφάλειας και άμυνας. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό στις συμβαστικές προτάσεις, όμως πραγματικά αυτό που ζητούμε είναι να συμπεριληφθεί η ανάγκη να έχουμε εστιακά σημεία όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τα δικαιώματα των γυναικών. Ιδίω σε ό,τι αφορά τι χώρε Αραβική Άνοιξη. Βέβαια, όχι μόνο, αλλά επειδή στην Αραβική Άνοιξη πολέμησαν, αγωνίστηκαν πολλέ γυναίκε που συμμετείχαν στι πορείε, στι διαμαρτυρίε, στι διαδηλώσει ε, που ήταν κατά των δικτατόρων και αυτό του ε, δημιούργησε προβλήματα και σε αυτέ αλλά και σε άλλε χώρε. Η ΕΕΔ και οι αντιπροσωπείε τη λοιπόν καλό θα είναι να έχει εστιακά σημεία focal points όπου οι γυναίκε ακτιβίστριε να ξέρουν ότι εκεί είναι ευπρόσδεκτε και μπορούν να συζητήσουν πράγματα και να έχουν και την υποστήριξη. Ελπίζω λοιπόν να την στήριξετε αυτή την πρόταση. Το ίδιο ισχύει για την τροπολογία 156 η οποία μιλά για το ότι κάθε ε, θα πρέπει να έχει έναν σύμβουλο για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Μπορεί να πηγαίνει λίγο μακριά, αλλά ε, όταν μιλάμε για ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τη ενέργεια, ιδίως σε αφρικανικές χώρες, αλλά και σε λατινοαμερικανικές ή ασιατικές χώρες. Αυτό ανησυχεί, ενδιαφέρει πάρα πολλούς πολίτες. Έχουμε πρόσφυγες, για λόγο, ε, πρόσφυγες λόγω του κλίματος. Ελπίζουμε λοιπόν να στηρίξετε, συνάδελφοι, την τροπολογία αυτή. Μια άλλη τροπολογία, η ασιατικες χωρες αυτο ανησυχει ενδιαφερει παρα πολλους πολιτες εχουμε προσφυγες για λογω του αφορά την δομή εργασίας μεταξύ ΕΙΕΔ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Working Structure, 160 τροπολογία. Νομίζω ότι είχαμε, είχαμε κάποια πρόοδο, είχαμε καλή συνεργασία με πολλούς από την ΕΙΕΔ και σε κάποιες από τις αντιπροσωπείες, αλλά όχι με όλες ακόμη τουλάχιστον. Όταν ζητάμε λοιπόν αποτελεσματική ροή επικοινωνίας πληροφοριών, μεταξύ Ευκομισιών, ε, Αντιπροσωπιών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει και θα βελτιώσει το έργο που επιτελούμε όλοι μας. Και κάτι άλλο που μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει της προσοχής που θα θέλαμε είναι ότι οι σχετικές μονάδες της ΕΕ, της Κομισιόν και των προσώπων θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τι απόψει και τι συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως αυτές εκφράζονται στα ψηφίσματά του. Και όχι μόνο αυτό, ε, αλλά και των Οργανισμών των Δικαιωμάτων και άλλων οργανισμών. Και θα πρέπει να μας αναφέρουν για το τι πρόοδο έχει επιτελεστεί σε σχέση με τις συστάσεις μας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θα βελτιώσει όχι μόνο τη συνεργασία αλλά και τα αποτελέσματα. Τέλος. Οι απόψει του Κοινοβουλίου που εκφράζονται στις εκθέσεις μας, στις συστάσεις μας, να εκπροσωπούνται, αν θέλετε, δεόντως ε, από μέλη της ΕΙΕΔ και από τις αντιπροσωπείες επαφές που έχουν με εξωματικούς τρίτων χωρών. Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης ε, πρέπει να ε, την χάνουν τη απαραίτητη υποστήριξης σε τρίτε χώρε. Ναι, μεν γίνεται, αλλά δεν είναι ακριβώ ομοιόμορφο το επίπεδο συνεργασία. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Εμεί θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία στο μέλλον με όλου. Θέλω λοιπόν να σα ευχαριστήσω και Λυπούμε, αλλά πρέπει να σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε σύντομα. to my Φεύγετε, πρέπει να ακούσετε την απάντησή μου. Για την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Εμείς προτείναμε ένα πολιτισμικό ε, ακόλουθο, κοινωνικό, α, ε, πώς σύμβουλο και ούτω καθεξής. Εντάξει, και μετά έχουμε μια γενική παρατήρηση. Ε, για, όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, αλλά ε, και τα τα πιέζουν. Και επίσης η ευρωπαϊκή πολιτιστική η πολιτισμική ταυτότητα που θέλουμε να δείξουμε προς τα έξω και αυτό είναι σημαντικό. Θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια γενική λοιπόν διατύπωση, δηλαδή ένα σύμβουλο, αλλά όχι απλά να λέει κλιματική αλλαγή για την κλιματική αλλαγή, να είναι και για άλλα θέματα, πολιτισμικά κτλ. Και βέβαια εξαρτάται και από τη χώρα. Τι πρόβλημα υπάρχει στην εκάστοτε περίπτωση. Ίσως στη Βραζιλία να έχουμε έναν εμπειρογνώμονα για το κλίμα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν είμαι σίγουρος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να είναι αποδοτικό από πλευράς ε, κόστους, ε, να το έχουμε κάπως υπό Το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό σκέλος της πρέσβειας δεν είναι ανεπτυγμένο όσο θα έπρεπε. Ε, ασχολούνται πιο πολύ με το εμπόριο και την ανάπτυξη. Και όπως είναι τα δημοσιονομικά μας αυτή τη στιγμή, καλό θα ήταν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η ευελιξία, ναι, αυτό θα το λάβουμε υπόψη μας. Ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη έχει κάνει μια πρόταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. έχει μια πρόταση, θα μα την εκθέσει πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά εγώ την υποστηρίζω και θα δούμε πώ μπορούμε να βρούμε μια λύση. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κρίσεων, εγώ δεν θέλω να έχουμε μια νέα διεύθυνση, directorate. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφόρων που έρχονται από διαφορετικά μέρη. Όχι να δημιουργηθεί μια νέα οντότητα, ένας νέος φορέας, ένα νέο τμήμα, διεύθυνση, όπω θέλετε πείτε το. Και το Συμβούλιο, Board, πάλι δεν λαμβάνει αποφάσεις. Τελικά είπατε εκπρόσωπο είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν σύμβουλοι που την συμβουλεύουν, ε, την βοηθούν να συντονίζει. Αν χρειαστεί και αν θέλει τη, στήριξη του Συμβουλίου, μπορεί να τη ζητήσει να την έχει, αλλά αυτή λαμβάνει τις αποφάσεις. Και αυτοί όλοι την συντονίζουν τη δουλειά της, την συμβουλεύουν. Και έχουμε και μια συμβαστική πρόταση του κ. Σαλαφράγκα. Ένα, στρατηγικό, ένα κέντρο στρατηγικού σχεδιασμού. Strategic Planning Center. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε γιατί ήδη υπάρχει. Ε, στην Helga Schmidt συγκεκριμένα. Πρέπει να βρούμε διαφορετική διατύπωση, αλλά διεύθυνση όχι. Με βρίσκει αντίθετο. Αυτά ως απάντηση. και τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε προβλήματα κάπου αλλού, εάν θέλετε. Θα ζητήσω από την Ανεμή τώρα. Ανεμή ναι, έτσι, από την άλλη να πάρει το λόγο. Ρομπέρτο, ε, ε, when you want to intervene... Ε. Και Ρομπέρτο, όταν θέλεις το λόγο, σήκω το χέρι και θα σου δίνουμε το λόγο αμέσως. Πρόεδρε, Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματο τη αντιπροσωπεία μου τους δύο εισηγητές για την εξωτερική δουλειά που κάναν και την καλή συνεργασία που είχαμε. Εκτιμώ ιδιαίτερα το πώς παλέψατε να ενσωματώσετε τις ανησυχίε ανησυχίες μας στις συμβαστικές τροπολογίες που σημαίνει ότι εν γέννη συμφωνούμε με το σχέδιο Υπάρχουν κάποιες μικρές ε, τροπολογίες, αλλά τίποτα το βασικό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας συγχαρώ εξ ονόματος της αντιπροσωπείας μου, την Βαρόνια Άστον και την ομάδα της, γιατί βοηθήσατε να βρεθεί συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κουσφοπεδίου. Ένα μείζον επίτευγμα και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της ίδιας, αλλά και των δύο πρωθυπουργών, που δείχνει τη χρησιμότητα των νέων δομών βέβαια. Αν μου επιτρέπετε ωστόσο, θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Υπάρχει μια τάση που το άκουσα και στην παρέμβαση της κυρίας Λούνετσεκ από τους πράσινους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπρόκ, ως κύριε Μπρόκ, σας μιλώ υπό την ιδιότητα του ως εισηγητή. Θα ήταν σκόπιμο να γράψετε ότι θα ήταν λάθος να πολλαπλασιαστούν ε, τα focal points ή διάφοροι έκτακτοι ειδικοί εκπρόσωποι, διότι θα καταλήξουμε τελικά να υπάρχει κόσμος που θα είναι πολλοί, αλλά θα δουλεύει μαζί. Δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο για μια ενοποιημένη προσέγγιση από πλευράς προσωπιών μας. Θα εγκρίνουμε λοιπόν το σχέδιο. Αυτά. Ευχαριστώ και πάλι ευχαριστώ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ. Δίκιο έχετε. Δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτό. Από τους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριο Τένοκ έχει ζητήσει τον λόγο. Ο κύριο Άτκιν. Όχι, ο κύριο Βαν Όντεν. Κάποια σχόλια. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι θέλουν αφενός να κάνουν πρεσβείες της αντιπροσωπείας. Μεταξύ αυτών και εσείς φαντάζομαι. Άλλοι δεν το πολύ πιστεύουν αυτό και σχετίζονται όλα αυτά βέβαια με την αντίληψη που έχουν για τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ιονή κρατικός ε, φορέας στη διεθνή σκηνή. Το να γίνει πρεσβεία ε, θα πρέπει βέβαια να έχουν και πλήρεις αρμοδιότητες ε, πρέσβεως με πολιτιστικές, αμυντικές ε, διαστάσεις. Θα αναγνωρίσετε ωστόσο πρόεδρες ότι πολλοί δεν το θέλουν. Για πολλούς λόγους και σε πολλά επίπεδα. Πολιτικά αφενός. Καταρχάς έχει αντίκτυπο στην έχει εκπροσώπηση των κρατών μελών. Υπάρχουν και χρηματοοικονομικές διαστάσεις η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική Βράση, εξορισμού, είναι πολυτέλεια και θα έλεγα εξορισμού επίσης και περιττή πολυτέλεια. Επιπλέον, όλες αυτές οι ιδέες των ε, διαφόρων για νέες αρμοδιότητες και μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν αν γίνουν περικοπές σε άλλους τομείς μπορεί από καιρού καιρού να είναι χρήσιμο να έχει 27 κράτη που συμφωνούν σε μια πρωτοβουλία ε, ενωσιακή θα μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμένο και όχι με τεράστιες διαστάσεις όπως μερικοί θέλουν να δείξουν. Ευχαριστώ. Να, περι... να απαντήσω σε όλους ακούγοντας πρώτα τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έκανα, υπέβαλα 10 τροπολογίες στην εκθεσή σας. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας. μεταξύ των οποίων και τη συμβιβαστική 13. Αν δείτε τα δύο κείμενα, κατά την άποψή μου η συμβαστική 13 δεν, δεν καλύπτει δική μου την 178, αφορά την γεωγραφική ισορροπία. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που ήδη ψηφίσαμε πριν από δύο-τρία χρόνια στο ψήφισμά μας τότε, όταν εξετάζαμε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική δράση και το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας. Η ερώτησή μου είναι πότε θα έχουμε τη θέση των εισηγητών για τις τροπολογίες. Η ψηφοφορία είναι αύριο και είναι πολύ βιαστική διαδικασία που δεν επιτρέπει σε όσους υπέβαλαν τροπολογίες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Δεν ξέρω αν έγινε συνάντηση των σκιωδών. Δηλαδή σήμερα συζητάμε, αύριο ψηφίζουμε. Πού είναι η διαφάνεια. Για την δική μου τροπολογία λοιπόν, δεν θεωρώ ότι 178 καλύπτεται από την δική σας 13 ε, συμβαστική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα γιατί ψηλό είχαμε σε μια μικρή αντιπαράτευση, αντιπαράτευση για ένα προηγούμενο θέμα γιατί είπα ότι ο συνάδελφός μου Τζέφρι Βαν Όρντεν δεν είναι ε, πάντοτε ορθολογικός. Ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι διαφωνούμε πάντοτε. Πάντως με, με, με τον ε, προηγούμενο ομιλητή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσουμε για την ΕΕ, αν λειτουργεί ή όχι. Εμείς πάντως έχουμε ανησυχίες και ιδίως ως προς το κόστος, αν είναι λογικό. Θα θυμάστε κύριε Πρόεδρε, όταν η υποεπιτροπή της Βουλής των Λόρδων ήρθε να πάρει κάποια συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής μας για το ζήτημα αυτό. Η έκθεση που δημοσίευσαν εν συνεχεία δεν ήταν τόσο εχθρική όσο θα την περίμενα εγώ ε, λόγω των μελών της υποεπιτροπής, γιατί είχαν πει και οι ίδιοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτούς το κόστος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου κάποιος που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορεί να είναι να μην είναι Βρετανός διπλωμάτης, αλλά είναι υψηλού επίπεδου δημοπλωμάτη, ε, να υποφελείται τελικά από αυτά τα οποία προσπαθούμε εμεί και ατομικά και συλλογικά να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω πάρα πολύ, απλά ε, εφιστώ λίγο την προσοχή του και του λέω ότι η πολιτική ε, και των συντηρητικό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως αγνωστικιστή, για να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά ε, τα υπέρ της ΕΕ. Δεν είναι και κάθετα, όμως αντίθετη. Συμφωνούμε πάντως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κόστος, κύριε Πρόεδρε, και αυτός θα πρέπει να είναι και ο γνώμονας που μας καθοδηγεί. Ευχαριστώ. Εγώ, μια και είμαι συντονιστή, θα μιλήσω επισήμω εξ ονόματο τη ομάδα. Δεν πρόκειται για τον τρίτο δρόμο. Ο μόνο τρόπο είναι, ο μόνο δρόμο είναι τη ECR. Και συνολικά, επειδή ήδη έχει λειτουργεί πλέον η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων κάποιο διάστημα, λοιπόν συνολικά την στηρίζουμε, ωστόσο θέλουμε να δούμε προστιθέμενη αξία ουδετερότητα ό,τι αφορά τον προπολογισμό και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των πόρων. Υπάρχει ένα αριθμό τομέων, για παράδειγμα, πρόσφατα στον διάλογο Πριστίνας Βελιγραδίου. Καθιάστον στήριξε τη διαδικασία αυτή. Μια χώρα μέλος δεν θα είχε επαρκή δυνατότητα να δώσει μια όθηση και στις δύο πλευρές. Οι Ιρανικές κυρώσεις επίσης βοηθούν πολύ στην αποτροπή της διάδοσης πυρηνικών όπλων. Πάλι 27 χώρες μέλη βαρύνουν περισσότερο από μία μόνη της ο αγώνας κατά της πειρατείας έξω από το κέρας της Αφρικής. Είχαμε εδώ τον πρόεδρο που καθόταν στη θέση σας και μας ευχαριστήσε για τη συνεργασία μας και δεν θα μπορούσε ποτέ να δράσει μια χώρα μόνη της, μια χώρα μέλος μόνη της. Άρα, συνολικά την δεχόμαστε. Ωστόσο, θεωρούμε ότι πρέπει να επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος κάθε μια χωρα ξεχωριστά, είτε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε είναι η Τσεχική Δημοκρατία, να ασκούν την διπλωματία τους ξεχωριστά. Και η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα πρέπει να προσφέρει κάποια καλύτερη προστιθέμενη αξία και ιδίω ό,τι αφορά τι εξοικονομήσει στα Υπουργεία Εξωτερικών του. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Δεν έχω δει ακόμα αρκετά στοιχεία που να μου δείχνουν ότι οι εθνικέ διοικήσει έχουν μειώσει το κόστο του. Παρατήρηση του κ. Βανόρδεν χωρί μικρόφωνο προ την κατεύθυνση του κ. Τάνοκ. Βεβαίω, κάθε κυβέρνηση θέλει εξοικονομήσει στον προϋπολογισμό της. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε καμία κυριαρχία. Απλώς θέλουμε να δούμε αν η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων... Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να απαντήσω στον ε, διπλανό μου. Η θέση μας πάντως, συνοψίζω, δεν είναι εχθρική. Είμαστε κάπως περισσότερο από απλά αγνωστικιστές, αν θέλετε, όπως το έθεσε ο Σερόμπερτ Μπερτάτκινς. Είμαστε, κλείνουμε μάλλον να είμαστε υπέρ, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ή τουλάχιστον αξία για τα χρήματα που δαπανούμε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στα θέματα που θέσατε και να δώσω και κάποιες λεπτομέρειες για τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνουμε. Για τα κυριότερα σημεία δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα όσα είπε ο Έλμαρ Μπροκ. Δηλαδή ότι αυτό που επιζητούμε είναι μια συνολική προσέγγιση. Δηλαδή να βάλουμε όλα μαζί τα θέματα εάν και να αποφύγουμε επικαλύψεις. Εάν πολλαπλασιάσουμε τις πτυχές, τις διαστάσεις, δεν εξοικονομούμε, αλλά πολλαπλασιάζουμε αυτά για τα οποία στην ουσία υποτίθεται ότι υπηρετεί, εξυπηρετεί η υπηρεσία εξωτερικών δάση. Για την σωστή δομή βέβαια προτείνουμε κάποιου συμβιβασμού. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιο όνομα στην δομή είναι ένα βήμα μπροστά. Στην κατεύθυνση που θέλουν να δουν οι πράσινοι. Δεν είναι ακριβώς η ίδια η πρόταση, εφού πρόκειται για συμβαστική πρόταση. Αλλά σώμαστε σαφώς υπέρ μιας δομής και υπέρ της οικοδόμησης, όπως λέει και η οδηγία, μιας συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Βρίσκω ότι είναι καλή η συμβαστική αυτή πρόταση, αν και δεν, είναι 100, δεν υπήρχε 100% την θέση των πράσινων βέβαια. χαίρομαι που βλέπω ότι η ομάδα των φιλελεύθερων είναι ικανοποιημένη με τη δουλειά μας. Ευχαριστώ και για τη συνεισφορά τους. Στην προφορική συμβαστική τροπολογία περιλαμβάνουμε και την αναφορά στην ρήτρα της γέφυρας καθώς και τη μελλοντική θέση της υπηρεσίας σε περίπτωση που οργανωθεί πάλι συνέλευση. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Σάριου Σουβόλσκη και βέβαια ο συμβασμός δεν απηχεί πλήρως τις τροπολογίες του διότι αλλιώς δεν θα ήταν απαραίτητο να γίνει να κατατεθεί συμβαστική τροπολογία, θα μπορούσαμε να βάλουμε τις δικές του. Πρόκειται συμβασμό, ωστόσο συμβασμό που περιλαμβάνει ένα κέριο στοιχείο δηλαδή την ανάγκη λήψης όλων των μέτρων για την εξασφάλιση της γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας. όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν που λαμβάνουμε από την τροπολογία σας. Βέβαια δεν παίρνουμε και το δεύτερο μέρος της τροπολογίας σας. Ακριβώς επειδή είναι συμβασμός. Νομίζω ότι είναι καλός συμβασμός, καλή συμβαστική τροπολογία και η οποία προσεγγίζει αυτά που λέτε εσείς. Εάν προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο θα διταχθεί η πλειοψηφία. Την πλειοψηφία εννοώ τώρα. Μπορεί να είναι τα πράγματα σε άλλη έκθεση υπό διαφορετικέ συνθήκε. Εδώ όμω πρόκειται για συμβιβασμό που νομίζω λαμβάνει υπόψη τι διαφορετικέ θέσει και ζητεί τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της γραφικής αντιπροσωπευτικότητα. Όπως είπε και ο κύριος Μπροκ προηγουμένως, προτείνουμε επίσης να λάβουμε μία παράθεση από την τροπολογία της κυρίας Μάριας Μίνιτς για τα ποσοστά στα διάφορα επίπεδα που δεν θέλουμε ωστόσο να ανατρέψουν την ισορροπία της εκθέσεως. Γι' αυτό μιλούμε για την περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα των γυναικών σε υψηλές θέσεις και την υπεραντιπροσώπευσή τους σε χαμηλές θέσεις. Προσπαθούμε στις συμβαστικές μας προτάσεις να συμπεριλάβουμε τις περισσότερες πτυχές από τις τροπολογίες των μελών. Υπάρχουν βέβαια θέματα ακόμη όπου σημειώνονται διαφωνίες και θα δούμε τι θα γίνουν ψηφοφορίες. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που λένε, που προτείνουν μάλλον πράγματα που αποφασίσαμε να μην τα βάλουμε σε τέτοιου είδους έκθεση για παράδειγμα, γίνεται διαπραγμάτευση για το χρηματοδοτικό. Πρέπει να το βάλουμε εκεί. Δεν είναι ένα θέμα προπολογισμού. Αλλά εδώ δεν είναι. Δεν μιλούμε για τον προπολογισμό της ΕΙΕΔ ουδέτερη ως προς τον προϋπολογισμό, αύξηση του προϋπολογισμού, μείωση του προϋπολογισμού. Δεν είναι το θέμα αυτό της έκθεσης αυτής. Πάντως και ο εκπρόσωπος της ομάδας των Βρετανών Συντηρητικών με τον ίδιο τρόπο μίλησε τώρα. Βέβαια έχουμε διαφορές στις προσεγγίσεις και ιδίω ό,τι αφορά το θέμα της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοσιονομικής αντιπροσωπευτικότητας, ό,τι αφορά τον προπολογισμό δηλαδή. Ε, ουδετερότητας, συγγνώμη, της δημοσιονομικής ουδετερότητας. Ευχαριστώ. Είπα ότι δεν είμαι ικανοποιημένο από την κάλυψη, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Το θέμα είναι σοβαρό. Στην έκθεσή σα πάμε πίσω σε σχέση με την παλαιότερη θέση του Κοινοβουλίου όπως είχε αποφασιστεί το 2010. Και εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο θα ήθελα να ξέρω γιατί. Και γιατί δεν έχουμε χρόνο και μηχανισμό συζήτησης. Σήμερα συζητούμε, αύριο ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για, οτιδήποτε, για οποιαδήποτε συζήτηση. Ούτε έγινε συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Ακολουθείτε μια ταχεία διαδικασία για να μην μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, κύριε Γκουαλτιέρη, και με την ε, αλλαγμένη διατύπωσή σας αλλάζετε την γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα με την γεωγραφική αντιπροσώπευση που είναι τελείως διαφορετικό. Λέμε για να καλυφθεί η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα της ΕΝΗΣ όπως απαιτεί το άρθρο 6.6 και 6.8 της απόφασης για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 8 Ιουνίου 2010 εισάγοντας συγκεκριμένα μέτρα για να, διορθωθούν, για να διορθούν οι γεωγραφικές ανισορροπίες που συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς να υπάρχει σωστή διόρθωση. Εγώ σας ε, παραθέτω δύο κείμενα. Ένα δεσμευτικό, το άρθρο 6 της απόφασης Συμβουλίου μετά την έκφραση της θέσης μας πριν από δύο χρόνια που λέει ότι η επιλογή θα γίνεται επί βάση την αξία εξασφαλίζοντας ε, γεωγραφική ισορροπία. Το προσωπικό θα εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη και η αναθεώρηση που προβλέπει το άρθρο 33.3, η αναθεώρηση που γίνεται τώρα δηλαδή, θα καλύπτει επίσης και το θέμα αυτό. Άρα εμείς περιμένουμε από εσά κυρία Άστον να το δείτε αυτό καθώς και προτάσεις όπως ενδικτεί, για, για μέτρα που μπορεί να καλύψουν πιθανές ανισορροπίες. Επιπρόσθετα ειδικά μέτρα. Το ίδιο αναφέρεται στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει στο σημείο 7 έχει την άποψη του Κοινοβούλιο, δηλαδή έχει την άποψη ότι επιπρόσθετα συγκεκριμένα μετά που περιλαμβάνεται στα άρθρα 6-6 του, Συμβουλίου, του Συμβουλίου για την ενίσχυση της γεωγραφικής και ισορροπίας και ισορροπίας φύλων θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα παρόμοια με τα αυτά που αναφέρονται στο, στην απόφαση Συμβουλίου 401 ε, του 2004. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε πρόοδο στην γεωγραφική ισορροπία και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Αυτό που αποφασίστηκε πριν από τρία χρόνια είναι ότι αν δεν υπάρξει διόρθωση θα υπάρξουν διορθωτικά μέτρα. Είναι προφανέ ότι εμεί ω Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσουμε τέτοια διορθωτικά μέτρα. Είδε μη, αλλάζουμε την πολιτική μα. Για το λόγο αυτό και έχοντας πλήρη επίγνωση του επίμαχου χαρακτήρα του θέματος, προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία αύριο για να έχουμε περισσότερο χρόνο για το θέμα αυτό. Για τις εκθέσεις σας κύριε Μπρόκ και κύριε Γκουαλτιέρη κάνετε πίσω σε σχέση με δεσμεύσεις που ήδη πετύχαμε και ε, παραχωρούμε και παραχωρούμε περισσότερα από αυτά που στην μέση του λόγου σας σας κατάλαβα, μετά μπερδεύτηκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα την δυνατότητα να δω κάποια στοιχεία σχετικά με <clears throat> το θέμα που έθιξε ο κ. Γκουαλτιέρη για την γεωγραφική ισορροπία. Μας δόθηκαν κάποια στοιχεία λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών για το 2010 και για φέτος. Τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν ωστόσο ότι έχουμε προσεγγίσει μια ισορροπία. 25% περίπου θα έπρεπε να προέρχονται από τις νέες χώρες μέλη. Γνωρίζω ότι αυτά όλα είναι καθαρά αριθμητικά στοιχεία και ότι η πραγματική ζωή είναι διαφορετική. Όμως η απόκληση από το μοντέλο που έχουμε υπόψη μας είναι ακόμα μακρύ, μα, μεγάλη. Τίθεται το ερώτημα τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Διαβάζοντας τώρα την έκθεση και στο άρθρο 35 βλέπω ότι μιλούν για εντατικοποίηση προσπαθειών για την καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και από την άποψη των φίλων και γεωγραφικά. Βεβαίως υπό λήψη υπόψη των αξιοκρατικών κριτηρίων. Γνωρίζουμε ότι τέτοιο εντατικό διάλογος υπήρξε ήδη το 2010 στην παρούσα Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί και στις τροπολογίες, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις. Τα δε στατιστικά αυτά στοιχεία τα οποία ευχαρίστω να σας δείξω, βλέπω ότι ο κύριος ε, Πέτεριν χαμογελά, αλλά δείχνουν τα στοιχεία αυτά και τη μεγάλη έλλειψη ισορροπίας. Εγώ αυτά τα σχόλια δεν τα λέω διόλου προσωπικά, τα λέω βεβαίως καθαρά αντικειμενικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να πω το εξής. Έχουμε ήδη συζητήσει για την έκθεση Gualtieri πρόκ, αλλά δεν ήσασταν παρόν, κύριε Βόλσκι. Δεύτερον, κάναμε και συνάντηση των σκιωδών εισηγητών την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως να μην είχατε προσκληθεί. Ε, αλλά δεν είχατε προσκληθεί ως σκιώδης, ίσως επειδή η σκιά σας είναι ευρύτατη. Έκανα, λέω, απαντά ο κ. έκανα συνάντηση με του Σκιώδη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είστε Σκιώδη ηγητή. Δεν είστε Σκιώδη ηγητή του Λαϊκού Κόμματο. Πέμπτη πρωί έγινε η συνάντηση των Σκιωδών. Όταν προσκαλώ τους Σκιώδη ηγητέ, μόνο αυτούς προσκαλώ και κανέναν άλλο. Πάτρικ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσουμε από ε, αυτού του θαυμάσιου σχεδίου εκθέσεως που έρχεται σε πολύ κατάλληλη στιγμή τώρα που η πάτη εκπρόσωπος ολοκληρώνει πλέον τον προβληματισμό της σχετικά με την αναθεώρηση που ως γνωρίζετε θα κατατεθεί μέσα στο καλοκαίρι Ιούνιο, Ιούλιο και γνωρίζω ότι η Πάτη εκπρόσωπος επιθυμεί να συζητήσει και βαθύτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο προχωρεί και ο δικός σας προβληματισμός. Νομίζω ότι η έκθεση θίγει πολλά σημαντικά θέματα και μπαίνει στην καρδιά των θεμάτων αυτών που μας απασχολούν και μας εσωτερικά. Το ρόλο και το καθεστώς των οργάνων διαχείρισης κρίσεων στην υπηρεσία μας, πώς να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερο στρατηγικό σκέπτεστε, πώς θα συνεργαζόμαστε με τα άλλα θεσμικά όργανα και βεβαίως ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης με ποιο τρόπο θα υποστηρίξουν περισσότερο οι αντιπροσωπείες μας το έργο των Ευρωβουλευτών όταν ταξιδεύουν απανταχού του κόσμου. Και χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα από τους βουλευτές σας ότι εκτιμούν το έργο που κάνουμε και ότι αυτό βελτιώνεται. Για τα σημεία επαφής, contact points ή focal points, και ιδίως λόγω των περιορισμένων μέσων που διαθέτουμε και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε και των προτεραιοτήτων διότι πρέπει να είναι εξοπλισμένες οι αντιπροσωπείες μας να μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις, προ... και τις πολιτικές προκλήσεις που ε, ε, βρίσκουν εκεί όπου βρίσκονται και να υπάρχουν πρόσωπα στα οποία να μπορείτε να απευθυνθείτε για θέματα, για παράδειγμα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων γυναικών κλπ. Αλλά και τον πολλαπλασιασμό των καθηκόντων που αν αυτά πολλαπλασιαστούν πάλι με τον αριθμό των 141, 141 αντιπροσωπιών θα γίνουν τελικώς πολύ δύσκολο να διαχειριστούν. Και με ένα τελευταίο σχόλιο, ίσως μπορώ να βοηθήσω την Επιτροπή σας για την γεωγραφική ισορροπία. όστα θα γνωρίζετε, μέγα μέρος του προσωπικού και επομένως και του προϋπολογισμού της ΕΙΕΔ μεταφέρθηκε αρχικώς από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου για ένα πλήθος ιστορικών λόγων και δυστυχώς οι συνάδελφοι των νέων χωρών μελών δυστυχώς υποεκπροσωπούνταν από τότε όμως νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει κάποια πρόοδο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια σε ό,τι αφορά την αύξηση της εκπροσώπησης των νέων χωρών μελών σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής μας. Το πιο πρόσφατο στοιχείο που διαθέτουμε είναι αν λάβουμε υπόψη και τους διορισμούς που επεξεργαζόμαστε τώρα, θα έχουμε 18% των αξιωματούχων μας κατηγορίας AD και 60% χαμηλότερων ε, βαθμών από τις νέες χώρες μέλη. Συγκρίνεται τώρα τα στοιχεία αυτά με τον συνολικό πληθυσμικό δυναμικό των νέων χωρών μελών θα δείτε ότι ναι, δεν υπάρχει ακόμη κάποιο έλλειμμα και σίγουρα θα χρειαστεί ε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και στη βάση των δεσμεύσεων της υπάτησης εκπροσώπου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ισοδίκαιη εκπροσώπηση όλων των χωρών μελών. Νομίζω ότι όμως αν μελετήσετε προσεκτικότερα τα στοιχεία θα δείτε ότι επιτελείται πρόοδος, υπάρχουν μια ή δύο χώρες μέλη εξ όσων εντάχθηκαν πρόσφατα αλλά υπάρχουν και που εκπροσωπούνται, αλλά και ορισμένες από τις πολύ παλιές χώρες μέλη. Η εκπροσώπησή τους δεν ισοδυναμεί με το πληθυσμιακό δυναμικό τους. Όπως είπα όμως, μας απασχολεί ακόμη και είπατε εκπρόσωπός μας έχει πει κατ' επανάληψη ότι αυτό που κυρίως μας απασχολεί είναι να προσελκύσουμε τους βέλτιστους και τους εφιέστατους αξιωματούχους. και η πρόταση που έχουμε επιτελέσει τελευταία νομίζω δείχνει ότι επιτελούμε πρόοδο και στην υλοποίηση της αρχής αυτής ικανοποιώντας ταυτόχρονα και το κριτήριο της γεωγραφικής αντιπροσώπευσης αλλά και της ισοδίκης αντιπροσώπευσης των φίλων. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας απευθύνω λίγα λόγια. Νομίζω το έργο της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου σε στήριξη της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο ίδιο πνεύμα. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για ορισμένους, σε ορισμένους εκ των ευρωβουλευτών σας που επένεσαν τα επιτεύγματα των προσπαθειών της υπάτης εκπροσώπου προσφάτως και εμά μας απασχολεί να δούμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε προς τη θέμενη αξία και στις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Είναι νεαρά ακόμη σε ηλικία η υπηρεσία μα, αλλά θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε και στα, όσα, μέσα στα πλαίσια των όσων προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Ο Ρομπέρτο και εγώ θα επανεξετάσουμε αυτό το θέμα της γεωγραφικής αντιπροσώπευσης Θεωρούμε ότι πάει καλά ωστόσο η εξέλιξη. Αλλά το θέμα αυτό δεν φύγει μοναχά τις ε, νέες χώρες μέλη. Και η Γερμανία υποεκπροσωπείται. Και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά που λέτε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο είναι να δούμε πού θα κάνουμε περικοπές. Ορισμένες χώρες μέλη απαιτούν να συμμετέχουν στην επιλογή και του αναπληρωτού εκπροσώπου στην κάθε αντιπροσωπεία. Θέλουν λοιπόν να επανεθνικοποιήσουν την υπηρεσία αυτή. Αλλά η μεταβατική φάση, η μεταβατική περίοδος έχει λήξει. Πρέπει η υπηρεσία αυτή να μπορέσει να διορίσει όπως γίνεται και με τους συνήθεις διαγωνισμούς, κονκούρ. Να μπορούν λοιπόν Πολωνοί νεαροί διπλωμάτες να συμμετάσχουν σε, αυτό, σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, στον διαγωνισμό. Και όμως έρχεσαι σε άλλη ε, τροπολογία σου αγαπητές Άριους και διαγράφεις τα θέματα αυτά. Ίσως διότι δεν έχεις κατανοήσει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ενώ αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να ξεπεραστεί και το, 100, και το 18%. Νομίζω ότι είναι η τροπολογία 178. Το αν θα λέει μέσα αντιπροσωπευτικότητα ή αντιπροσώπευση, αυτό νομίζω ότι είναι λιγότερο σημαντικό. Πρόκειται για, ε, μιλούμε για το άρθρο 6 και το άρθρο 6.8 και εκεί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, όπως επίσης και για την ισοδίκη και την προσώπευση των φύλων όπως είπα και προηγουμένως. Νομίζω ότι μάλλον θα τα καταφέρουμε. Για το θέμα αυτό, ωστόσο, μας δήλωσαν την πλήρη υποστήριξή τους όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και της δικής σου ομάδας. Έτσι έχει κατάσταση. Νομίζω ότι, ωστόσο, με λίγες κονδυλιές θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Αλλά σε τέτοια έκθεση δεν είναι δυνατόν να υπερασπίζεται κανείς λησαλέα και την τελευταία του λέξη και την τελευταία του λέξη σε κάθε τροπολογία. Όλοι θα κάνουν κάποιες παραχωρήσεις ώστε να υπάρξει στο τέλος μια, να διατυπωθεί και να συνταχθεί στο τέλος μια λογική συνεκτική πρόταση. για τα, θέματα που για τα θέματα που έθεσαν οι Βρετανοί συνάδελφοι. Βεβαίως οι χώρες μέλη είναι κυρίαρχε, είναι όμως και συμβατικώ υποχρεωμένε. δεσμεύονται συμβατικά να υλοποιήσουν τα όσα έχουν υπογράψει. Πρόκειται για πρωτογενέ δίκαιο. Άρα έτσι πρέπει να γίνει. Έγινε και μια προσπάθεια να το συνδυάσουν κάποιοι εδώ και με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να διασφαλίζεται, λέει, διαβάζω μια τροπολογία, κάθε αντιπροσωπεία να διαθέτει την τεχνογνωσία στη συγκεκριμένη χώρα για τα θέματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη χώρα. Και σε παρένθεση λέει μέσα κλιματική αλλαγή, κοινωνικά δικαιώματα, συνδικαλιστικά κλπ. Αυτά όμως δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόσωπο σε κάθε αντιπροσωπεία για κάθε ξεχωριστό τέτοιο θέμα. Μπορεί ένα να έχει τεχνογνωσία για πλοίο από τα θέματα αυτά. Αν μπορέσει να βρεθεί μια τέτοια συμβαστική λύση, τότε πολύ ευχαρίστω. Θα ήθελα να ακούσω τι απόψει σα. Ρομπέρτο, εσείς τι νομίζετε. Really, I have nothing particular. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα το ξανασκεφτούμε πώς θα διατυπώσουμε αυτό το κείμενο της συμβαστικής τροπολογίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ της αντιπροσωπευτικότητας και της αντιπροσώπευσης. Στην ουσία μιλάμε για όλα τα αναγκαία μέτρα αποκατάσταση. Αυτό είναι το ουσιαστικό παραθέτουμε και την απόφαση του Συμβουλίου. Η διατύπωση νομίζω είναι καλή. Τώρα να δούμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν έχω να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μετρήσαμε τον πληθυσμό με το σωστό τρόπο. Σε 12 κράτη, τα 12 κράτη, νέα κράτη έχουν 19,5% του πληθυσμού της Ένωσης και τα 18% των διπλωματών. Όχι, αν χρησιμοποιήσουμε τις... Οι 12 χώρες η βασική ε, τιμή αναφοράς δεν είναι μόνο ο πληθυσμός και κατά βάση θα έπρεπε με βάση την σωστή αυτή ε, μερίδα αναφοράς το 26% θα πρέπει να είναι. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή ποιος είναι αυτός ο τρόπος υπολογισμού που μιλάτε. Δεν μπορείς να τον παρακολουθήσω. Τέλος πάντων. Προχωράει πάντως η κατάσταση και κάνουμε περισσότερα στην έκθεση αυτή. Ζητάμε να προχωρήσει περαιτέρω. Συμφωνούμε επ' αυτού. Το θέμα είναι η διατύπωση, δεν η στάση. Ευχαριστώ. Νομίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ελπίζουμε να έχουμε ευρεία συνένεση αύριο. Για να υπάρξει αντίκτυπος στις περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστώ. diesem uh, Frau Nates, wir haben noch eine Stellungnahme, die Sie darzustellen haben. Ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και καταπολέμηση των απατών. Η κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αντικαθιστώ την Ρενάτε Βέμπερ που ήταν η στάκταρ της γνωμοδότησης αλλά είναι και επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικής Παρατήρησης στην ε, Ουρουάη. Με παρακάλεσε λοιπόν να την αντικαταστήσω, να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή της και βέβαια δέχτηκα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, εξ ονόματος θα ήθελα να πω τα εξής. Όπως επισημαίνει, υπάρχει σημαντική βελτίωση το 2011 σε ό,τι αφορά την ανάκτηση πόρων και μη μάλλον και αχρήστους καταβληθέντων ποσών, όπως σε ό,τι αφορά προ πρωταξιακά κονδύλια. Επίσης έχουμε το σχέδιο πολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αλκοόλ και στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης. Σημαντικό συμπεριλαμβάνονται επίσης διατάξεις κατά της απάτης σε νέε ή αναδιαπραγματευόμενε συμφωνίε διμερεί. Χαιρετίζει η Ένωση επίση ε, η γνωμοδότηση, ε, την αναδιάργανωση τη Όλαφ. Έχουμε πλέον κάποιε διοικητικέ διευθετήσει και με τρίτε χώρε και κάποιου διεθνού οργανισμού για την ενίσχυση τη δυνατότητα Όλαφ να αντιμετωπίζει την απάτη σε τομεί που εντάσσεται στη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Επίσης, ζητεί γνωμοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ε, και κατάλληλη δαπάνη των προλαμβάνοντα υπόψη τα πορίσματα της ετήσιας έκδοσης του Ανακτικού Συνεδρίου για την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάποια ασφάλματα δεν ανοιχνεύτηκαν μέσω των ελέγχων της Κομισιόν. Άλλες συστάσεις προτείνει η συγκήτρια να συμπεριληφθούν οι διατάξεις καταπολέμησης της απάτης όλες τις δημερείς συμφωνίες με τις χώρες και να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την παράταση της εντολής των αποστολών της Ένωσης. Και αυτό για να υπάρξει αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση των πόρων. Η συγγήτρια κατέθεσε τρεις τροπολογίες, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στην ανάγκη βελτίωσης της χρηματοδότησης για τις αρχές νόμου και στα κράτη-μέλη και στις γειτονικές χώρες με στόχο την καλύτερη προστασία των χρηματοπιστωτικών συμφέροντων της Ένωσης. Οι τροπολογίες των συναδέλφων επίσης, σίγουρα θα συνεισφέρουν σημαντικά στην έκθεση, όπως όσε αφορούν το διασυνορικό χαρακτήρα της απάτης, συμπερίληψη διατάξεων καταπολέμησης της απάτης ε, στα προγράμματα δαπάνη στο πλαίσιο του νέου πολιετού δημοσιομικού πλαισίου, όπως και η ανάγκη εντατικοποίησης της ε, τελωνιακής απάτης. Η συνάδελφος Βέμπερ έχει εκφράσει κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Τροπολογία του Μίχαλ Γκάλερ, αριθμόν συγκεκριμένα. Η Ρενάτε Βέμπερ προτείνει ψηφοφορία κατά τμήματα για την τροπολογία αυτή. Ο λόγος είναι ότι πιστεύει πως το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας Γκάλερ επισημαίνει την Κροατία και την ε, Μακεδονία ε, αστόχους. Και ζητά επίσης η κυρία Βέμπερ βηματική ψηφοφορία στην τροπολογία 9 της κυρίας Φλάσκο Βαμπένοβα. Ή μάλλον όχι λέει να καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία, διότι πιστεύει ότι ναι μεν οι κίνδυνοι για την υγεία που αναφέρονται εδώ ισχύουν, αλλά δεν είναι και το βασικό αντικείμενο αυτής της γνωμοδότησης. Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Η συνάδελφος Ρενάτε Βέμπερ προσπάθησε να εκφράσει με το σχέδιο γνωμοδότησής το οποίο σας ε, υποβάλλει προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm taking... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ του Μίχαλ Γκάλερ που είναι ο σκιώδης συζητήτη ε, για το ΕΛΚ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί και ο ίδιος είναι σε μια αποστολή στο εξωτερικό εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη συντάκτρα της γνωμοδότησης κυρία Ρενάτε Βέμπερ για την καλή της δουλειά. Το σχέδιο γνωμοδότησής της καλύπτει πολλές σημαντικές πτυχές που θα πρέπει ε, να εκφράζει σχετικά τις απόψεις της ΙΑΦΕΤ. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις τροπολογιών που ουσιαστικά αποτελούν προσθήκη για να τονιστούν κάποιες πτυχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα ότι η συγγήτρια ήδη ε, αντέδρασε στην ε, τροπολογία 1 επί της παραγράφου 1 Βέβαια έχουμε πέντε τροπολογίες συνολικά. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο να μου επιτρέψει να μιλήσω για αυτές τις τροπολογίες. Τώρα έχουμε στην τροπολογία 2 την παράγραφο 2. Το ελληνικό συνέδριο θεώρησε ότι ο ελεγκτικό μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικό και αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να επιτύχει βελτιώσει ακολουθώντα τι συστάσει ακριβώ αυτέ του ελεγκτικού ε, συνεδρίου αλλά και την άποψή μα ε, περί τη απαλλαγή. Τροπολογία 3 για την παράγραφο 3. Εν ώψη του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου το 2014-2020 ε, θα πρέπει οι προσπάθειες για τη βελτίωση των διατάξεων κατά της απάτης να βελτιωθούν και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αποτροπή ε, καταχρήσεων και στα κρατημέλη και σε τρίτες χώρες. Ε, τροπολογία 4 παράγραφο 5 για διμερείς, πολυμερείς ε, συμφωνίες με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να υπάρξει μια τυπική πρότυπη ρήτρα για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία θα αναπτυχθεί και θα συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες. Τροπολογία 5, παράγραφο 6. Εκεί ε, σε ό,τι αφορά τις δικασίες διαγωνισμού δημοσίων προμηθειών βλέπουμε κάποιες αδυναμίες. Αυτές θα πρέπει να διορθωθούν πάρα πολύ σύντομα. Σε αυτόν τον οργανισμό τον τόσο νέο, την ΕΕΔ δηλαδή, είναι καλό να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας και να θεσπιστούν από την αρχή καλές πρακτικές. Ο Μιχαήλ Γκάλερ ελπίζει ότι οι συνάδελφοι μπορούν να στηρίξουν τις προτάσεις αυτές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την συνάδελφο Πιμαλάκη που λείπει υποστηρίζει την γνωμοδότηση. Οι τροπολογίες έχουν στόχο να βελτιώσουν σε κάποιες μικρές ε, διαφοροποιήσεις το κείμενο υπογραμμίζεται η ανάγκη καταπολέμησης ε, της απάτη που σχετίζεται με τις τελωνιακές δραστηριότητες, απάτη που διαπράτεται όλο ένα και περισσότερο διασυνοριακά και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ισχυρό, ισχυρή δέσμευση από πλευράς εταίρων χωρών. Επίσης καλωσορίζει την πρωτοβουλία βελτίωσης της ικανότητας αντιμετώπισης ε, της απάτης με την ενίσχυση της ΟΛΑΦ και προσβλέπει στην γρήγορη ολοκλήρωση της υφιστάμενης νομοθετικής διαδικασίας για την αναθεώρηση του ψηφίσματος του 99 που θα δώσει το πλαίσιο που χρειάζεται για να υπάρχει μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αυτά. η εκπρόσωπος της ηγήτριας. Είδα, ήδη σας ανέφερα πολλές τροπολογίες και ανέφερα ε, ποιες μπορούμε να δεχθούμε και ποιες όχι. Μία από αυτή είναι η τροπολογία 2. Εδώ ζητάμε να υπάρξει ψηφοφορία κατά τμήματα στην τροπολογία 1 του συναδέλφου Γκάλερ που δεν υποστηρίζουμε την προσθήκη που θέλει να βάλει στην παράγραφο αυτό ο κύριος Γκάλερ. Πιστεύω ότι αν κατάλαβα καλά από το σημείωμα θα υποστηρίξουμε τις περισσότερες από τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση. Στις 27 Μαΐου θα έρθει ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ουκραϊ της Ουκρανίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας και ο Βουκ Κέρεμεκ, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο εκείνη την μέρα θα έρθουν. Συνάντηση όμως τότε δεν έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε μια εκτακτή συνάντηση τότε για να συζητήσουμε τους δύο αυτούς ανθρώπους ή όχι. Υπάρχει αντίρρηση. Μπορώ να ρωτήσω και του συντονιστέ, αλλά τέλο πάντων εγώ αυτό προτείνω. Δεύτερον, Θέλετε να σας στείλω εγγράφο στην έκθεσή μου για τη Βραζιλία ή θέλω να σας το πω προφορικά. Εσένα δεν σε νοιάζει γιατί ήσουν εκεί. Μια χαρά είναι το εγγράφος, πρόεδρε. Μια παρατήρηση πάντως προφορικά. Θέλει περισσότερη δουλειά η Λατινική Αμερική. Όχι γιατί η Βραζιλία είναι στους BRIC, αλλά και για άλλους λόγους. Είναι σημαντική. Όχι μόνο οικονομικά, στρατηγικά Ο κ. Μίλαν Μόν ήταν εκεί και διαπιστώσαμε και φοβερό ενδιαφέρον και πολλές παρανοήσεις. Πρέπει να έχουμε μόνιμη, πιο συχνή συζήτηση μαζί τους. Και τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα της Βραζιλίας ήθελαν με πάθος να συζητούν μαζί μας. Θα έρθουν κάποιοι το Μάιο και πραγματικά πρέπει να μιλά μαζί τους περισσότερο η Ευρώπη. Κύριο Στένοκ, συμφωνώ να κάνουμε περισσότερα για τη Λατινική Αμερική. Άρα είναι κρίμα που είναι τμήμα των BRICS η Βραζιλία, είναι η τοπική υπερδύναμη και δεν κάνει τίποτα στην αυξήση αυξήσει την αντιπροσωπεία της εδώ. 14 χρόνια είμαι στο κοινοβούλιο, ένα Βραζιλιάνο δεν είδα, Κολομβιανούς, Χιλιανούς είδα, έρχονται, είναι δραστήριοι. Η Βραζιλία είναι ένας υπνότων γίγας. Και εγώ και μιλάω και βραζιλιάνικα, μια χαρά και δεν έχω βρει κανένα να το κουβεντιάσω. Προφανώς επειδή δεν ξέρουν ότι μιλάει τόσο ωραία από το γαλλικά ο κύριος Τάνοκ. Γι' αυτό δεν έρχονται. Γιατί πιστεύω ότι η βραζιλιανική πρεσβεία προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μας. Προφανώς ε, πηγαίνουν στους συναδέλφου που είναι σε επιτροπέ που έχουν σχέση μαζί τους. Του Μερκοσούρ για παράδειγμα. Ε, γι' αυτό είναι σημαντική η αντιπροσωπεία. Ήταν η πρώτη φορά που στείλαμε αντιπροσωπεία στη Βραζιλία για πολιτικέ διαβουλεύσει και όπω ανέφερε ο πρόεδρο Μπρόκ, εκτίμησε ιδιαίτερα την επίσκεψή μα αυτή. Ε, διαφάνει ανάγκη διαβουλεύσεων γιατί υπήρχαν τόσε παρανοήσεις και η επικοινωνία μαζί τους μας επέτρεπε να καταπολεμήσουμε αυτές τις παρανοήσεις. Πιστεύω ότι ήταν ενδεικτικό το πόσο σημαντική τόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στην επίσκεψή μας. Σχεδόν τους πάντες είδαμε, μόνο την πρόεδρο δεν είδαμε. Και αυτό είναι δείγμα της σημασίας που έδωσαν στις διαβουλεύσεις. Πολύ ωραία τα είπε ο πρόεδρος Μπροκ, πολύ ωραία προείδευε. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε μια πολύ πιο καλή σχέση. Όπως το τόνισε και ο Τσάρλς. Συμφωνώ με την αξιολόγη, με την εκτίμησή σας ότι παίζει σημαντικό ρόλο η Λατινική Αμερική. Εγώ θέλω να προτείνω κάτι, πρόεδρε μόλις υπάρξει η γραπτή σας έκθεση, να κάνουμε μια συζήτηση για την έκθεση που θα μας δώσει την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εκ των, υστέρων, εκ των ε, προτέρων και να οργανώσουμε συζήτηση. Η Βραζιλία και η Ελληνική Αμερική παίζει ρόλο και για τις ε, πρόσφατες αλλαγές στη Βενεζουέλα και για τις πρόσφατες αλλαγές στην Ουρουγουάη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπατε. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Πρώτη φορά που πήγε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στην ε, Βραζιλία. Συμφωνώ ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις Χρειάζονται αρκετέ διευκρινήσει. Ο διάλογο αυτό λοιπόν δείχνει μια αλλαγή ρότας. Εμφανίζεται η επίγνωση της ανάγκης διαλόγου και θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο με τους Βασιλιανούς. Να έχουμε μια πιο south-south προσέγγιση ιδίω για να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσεις. Ευχαριστώ. Με αυτή σα την παρατήρηση θα μιλήσω αγγλικά. Υπήρχε η συμφωνία μεταξύ Προέδρου Λούλα και εμού. Είμαστε τα βαρέα βάρη στον ε, παγκόσμιο τελικό της Βραζιλίας, αν καταλάβατε τι εννοώ. Πάντως η Βραζιλία δεν θέλουν τόσο πολύ να είναι ενταγμένοι σε αυτά τα BRICS. Ακόμη κάπως τους ανησυχεί το βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών η οι γκρίνγκο που είναι προς βοράν. Θέλουν συνεργασία με την Ευρώπη και γι' αυτό αυτή η πρόταση για μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών Μερκοσούρ με την Ευρώπη. Η Αργεντινή ίσως οδεύει προς την επόμενη πτώχευση η κατάσταση είναι δύσκολη επίσης στην ε, Παραγουάη. Η Βενεζουέλα ίσως θέλει να αναλάβει τα Ινία. Ε, Αλλά διαμορφώνεται μια νέα σκακέρα συμφερόντων που πρέπει να λάβουμε υπόψη και γι' αυτό αγαπητέ Charles θεωρώ ότι θα έχουν και περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε αύριο. Και ε, πάλι ελπίζω να βουτυχτούμε σε συμβασμού. Όχι, habe das alles durcheinander, ja.